ένα, δύο, τρία. Υπότιτλοι είναι ευχαρίστηση κύριε Παπανδρέου να σας υποδέχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που δεχτήκατε την ε, πρόσκλησή μας να συνεισφέρετε σε μία από τις ακροάσεις μας στην Επιτροπή για την κρίση. Γνωρίζουμε βεβαίως ε, τα στοιχεία του βιογραφικού σας, δεν θα το διαβάσω τώρα ολόκληρο, αλλά έχετε παίξει σημαντικό ρόλο στην ελληνική πολιτική η επί σειρά ετών, είτε στην αντιπολίτευση, είτε στην κυβέρνηση, είτε τώρα ως Πρωθυπουργός και βεβαίως ε, είναι σημαντική η συνεισφορά σας. Όπως όλοι ξέρουμε υποφέρεται αυτή τη στιγμή ε, λόγω της κερδοσκοπίας κατά της Ευρωζώνης και της Ελλάδας ιδιαίτερα. Η κατάσταση δείχνει πως η εμπιστοσύνη στο ευρώ δεν έχει ακόμα εδραιωθεί 100%. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και το πώς θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση το ευρώ αποδείχτηκε στην αρχή βράχο σταθερότητα στην ε, οικονομική κρίση και χωρίς αυτό πολλά κράτη-μέλη θα ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι τώρα. Τα μέλη της Ευρωζώνης αποφάσισαν την τρίτη που μας πέρασε να σας στηρίξουν στην περίπτωση που θα ζητήσετε βεβαίω αυτή τη στήριξη. Μέχρι στιγμή δεν το έχετε κάνει. Γνωρίζω πω ο Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Παπακουσταντίνου, ζήτησε, όπω είπε, ένα όπλο να είναι πάνω στο τραπέζι. Και είπε πω υπάρχει αυτό το γεμάτο όπλο πάνω στο τραπέζι, οπότε αν το χρειαστώ θα το χρησιμοποιήσω και αυτό είναι καλό. Θαυμάζω το θάρρο σα, κύριε Πρωθυπουργέ, για τα μέτρα αυτά τα φιλόδοξα, τα οποία αποτελούν πάρα πολύ πρόκληση όσον αφορά τις οικονομίες και την λιτότητα και αυτή τη στιγμή πληρώνουμε το γεγονός ότι τα πρώτα χρόνια της Ευρωζώνης κάποιες χώρες και η δική μου, η Γερμανία και η Γαλλία και άλλες δεν σεβάστηκαν τα κριτήρια σταθερότητας όπως αυτά είχαν οριστεί. Γι' αυτό νομίζω πως είναι σημαντικό να αποδείξουμε τώρα πως ακόμη και σε καιρούς δύσκολους μπορούμε να ξαναβρούμε το δρόμο προς την ομαλότητα. Πρέπει να προσθέσω μια τελευταία λέξη. Είμαστε όχι μόνο κατάπληκτη, αλλά σοκαρισμένοι από το ότι αυτές οι τράπεζε και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πριν από λίγους μήνες ήταν ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία και διασώθηκαν με τα χρήματα του φορολογημένου, χρησιμοποιούν την πρώτη ευκαιρία που βρίσκουν για να κερδοσκοπήσουν κατά του ευρώ. Και βεβαίω να βγάλουν χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Και βεβαίω ε, δεν θα εκπλαγείτε πως όταν θα ρυθμίσει τα παράγωγα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβει σκληρά μέτρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο, σας καλωσορίζουμε και πάλι σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κλίντς, ε, κυρίες και κύριοι. Είναι πάντα μεγάλη μου τιμή να απευθύνομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τους τελευταίους πέντε μήνες από όταν εξελέγην έχω παρευρεθεί σε διάφορα πάνελ, έχω δώσει συνεντεύξεις, ε, διασκέψεις, αλλά είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα καθώς ε, δεν απευθύνομαι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά σε αυτό το οποίο θα λέγω εγώ το σημαντικότερο θεσμικό όργανο δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει σημαντικό ρόλο να παίξει και μπορώ να πω πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συχνά είναι μπροστά ακόμη και από το έργο των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων αντιμετωπίζει τα πολλά ζητήματα που έχει μπροστά της η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην ε, ολοκλήρωση που αφορά βέβαια και την διεύρυνση αλλά και την εμβάθυνση των θεσμών μας. Παλέψαμε και εγώ προσωπικά υπό την ιδιότητά μου ε, υπουργό Εξωτερικών και επί της ε, Προεδρίας όταν μιλούσαμε για το λεγόμενο Σύνταγμα που αργότερα έγινε η Συνθήκη της Λισαβόνας για να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και νομίζω πως ε, το σώμα θα καταστεί ένα σημαντικός παράγοντας ε, λήψης αποφάσεων που θα προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών μας. Και βεβαίως μια τέτοια πρωτοβουλία είναι η δημιουργία της ε, δικής σας Επιτροπής για την οικονομική, δημοσιονομική και κοινωνική, όπως πολύ σωστά είπατε, κρίση. Πώς θα όριζα εγώ την κρίση. Πρώτα απ' όλα, για να δούμε τα πράγματα λίγο γενικότερα, είναι μια κρίση παγκόσμιας διακυβέρνησης, παγκόσμιας δημοκρατικής διακυβέρνησης και όταν πανηγυρίζαμε για το τέλος του ψυχρού πολέμου δεν είδαμε ότι η ιστορία τελικά δεν τελείωσε, προβλήματα ακόμα υπήρχαν και καθώς οι κρατικοί μηχανισμοί του πρώην Ανατολικού Μπλοκ κατέρεαν, γίναμε πάρα πολύ δογματικοί στην πίστη μας στις ε, δυνάμεις της αγοράς. Και είχαμε δημιουργήσει έναν ε, νέο άρχοντα της ε, αγορές χωρίς καμία ρυθμισή και πίσω από αυτές υπήρχαν κάποιες δυνάμεις ε, που πολύ συχνά έλεγχαν τις αγορές και την πολιτική μας και αυτό είδαμε με την κρίση πριν από δύο χρόνια το γεγονός ότι υπήρχε έλλειψη διαφάνειας ότι πίσω από την λεγόμενη αυτή καινοτομία είχαμε σχήματα που μπορούσαν να αποφύγουν οποιοδήποτε είδους έλεγχο, οι βέλτιστες πρακτικές, δημιουργούσαν φούσκες και οι φούσκες αυτές πληρώθηκαν. Δυστυχώς από τους πολίτες μας, σε όλο τον κόσμο και από αυτούς που δεν είχαν καθόλου ευθύνη ή είχαν ελάχιστη ευθύνη. Νομίζω πως είναι μεγάλη η πρόκληση και αυτή τη στιγμή οι πολίτες μας αισθάνονται πως εμείς, ε, η διεθνής κοινότητα, δύο χρόνια από όταν ξεκίνησε η κρίση, αν και σιγά σιγά την ξεπερνάμε, δεν καταφέραμε να κάνουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Και αυτή είναι μια μεγάλη ε, πρόκληση και αυτό δείχνει την και δίνει μια αίσθηση αδυναμίας, μια πολύ επικίνδυνη αίσθηση, γιατί αν χάσουν οι πολίτες μας την ε, εμπιστοσύνη τους στην αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων, των θεσμών σε εθνικό ή διεθνές ή ευρωπαϊκό επίπεδο θα αναζητήσουν άλλες μεθόδους, λαϊκισμό, βία, φονταμεταλισμό, ακραίες τάσεις, πόλωση, αυτό θα δούμε στις κοινωνίες μας, ανά τον κόσμο. Οπότε πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα πρέπει και πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια είναι ένα μάθημα εν τη καθώς ε, έχουμε θεσμικά όργανα που κυβερνούν μια ευρύτερη περιοχή με τους ε, κανόνες εκείνους ε, και την κοινή εκείνη κυριαρχία που μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα για την οικονομία μας, την παγκοσμιοποιημένη, αλλά και για άλλα ζητήματα. Ζητήματα όπως κλιματική αλλαγή, ζητήματα όπως η αντιμετώπιση της μετανάστευσης, της στόχιας κτλ. Οπότε εγώ θα έλεγα να μην επιστρέψουμε στα ίδια όπως παλιά και χαίρομαι που το συζητάτε στην Επιτροπή σας. Το τιμμα είναι υψηλό, το τιμμα αυτή τη στιγμή είναι υψηλή ανεργία, μειωμένη μισθή και ένα μέλλον το οποίο πιθανώς ε, είναι δυσμενές. Πρέπει λοιπόν να αποστείλουμε ένα ισχυρό, ισχυρό μήνυμα στην επόμενη συνάντηση των G20 όπου συμμετέχουν αρκετά κράτη-μέλη της Ένωσης. Είναι μια ευκαιρία για να προωθήσουμε ένα πρόγραμμα των κανονισμών εκείνων που θα θέλαμε εμείς να δούμε. Εγώ στις ε, πολλές ε, συναντήσεις μου τις τελευταίες εβδομάδες με πολλούς ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση συναντήθηκα με τον Γκόρντον Μπράουν στο Λονδίνο, με τον Χωσέ Λουίς Σαπατέρο, πήγα στο Βερολίνο, μίλησα με την Αγγέλα Μέρκελ, στο Παρίσι με τον Νικόλα Σαρκοζή, με τον Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, τον επικεφαλής του Eurogroup και προέκυψε από αυτά και μια πρωτοβουλία που αφορούσε τα credit default swaps, όπως λέγονται, τις συμφωνίες ανταλλαγής κινδυνοθέτησης. Αυτά τα Συζήτησα και την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα στη ΣΥΠΑ και του ζήτησα εκ μέρους ημών πιο στεναρή λήψη αποφάσεων ε, στον τομέα της ρύθμισης σε διεθνές επίπεδο και χάρηκα για το ότι η απάντηση ήταν θετική. Βεβαίως καμιά φορά διάβολος κρύβεται τις λεπτομέρειες αλλά προφανώς ε, το γεγονό ότι αυτό το αντιλαμβάνω σε υψηλότερα επίπεδα ΣΥΠΑ είναι ένα θετικό σημάδι. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με την Ελλάδα. Είμαστε στο κέντρο μια ε, οξία και περίπλοκη ε, κρίση που έχει προκληθεί πρώτα απ' όλα από εσωτερικά διαρθρωτικά προβλήματα, τα οποία όμω μετά οξύνθηκαν από παγκόσμια δημοσιονομικά προβλήματα από την κρίση και όπως είπατε κύριε Πρόεδρε από την έντονη πίεση της κερδοσκοπίας, της κερδοσκοπικής κερδοσκοπίας. Θα ήθελα να είμαι σαφής. Δεν αναζητώ αυτή τη στιγμή από διοπομπαίο τράγο. Δεν προσπαθώ να ρίξω τις ευθύνες σε κάποιον άλλον. Πρώτος αναγνώρισα πως είναι ευθύνη της χώρας μας να αντιμετωπίσουμε τα διαρθρωτικά μας προβλήματα. Είναι δική μας ευθύνη να διορθώσουμε λάθη που εξασθένησαν τη θέση της Ελλάδας και μάλιστα στη μέση μιας παγκόσμιας δημοσιονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα ενώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διορθώσουμε αυτά τα λάθη που κληρονομήσαμε. Είναι παράδοξο και το αναφέρατε πως ε, η μοίρα μας κρίνεται από αυτούς, από τις ίδιες δυνάμεις, είτε είναι στην αγορά των Συμφωνίων Ανταλλαγής Κινδυνοθέτησης ή των εταιριών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δεν αναγνώρισαν τα λάθη του παγκοσμίου ε, συστήματος και ήταν υπεύθυνοι για τα ελαττώματα αυτά, γιατί δεν, υπήρχε, δεν τα επιτήρησαν σωστά και σήμερα εμείς πληρώνουμε γιατί μας επιτηρούν, ενώ εμείς τους γλιτώσαμε. Είναι παράδοξο λοιπόν, οι φόροι των λαών μας γλίτωσαν αυτές τις τράπεζες και όμως τώρα μας χτυπάνε για το έλλειμμα που δημιουργήσαμε για να τους γλιτώσουμε. Και οι λαοί μας τα πληρώνουν αυτά. Και αυτό είναι το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να τονίσω. Ναι, γνωρίζω πως η Ελλάδα έχει διαρθρωτικά προβλήματα, αλλά υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα που πρέπει να δούμε. Το πώς θα δημιουργήσουμε τα απαραίτητα βήματα για να προστατεύσουμε τις απαραίτητες αλλαγές που κάνουμε. Να σας πω λοιπόν το τι κάνουμε, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η κυβέρνησή μας ανέλαβε πριν από πέντε μήνες με μια ισχυρή εντολή για αλλαγή. Οπότε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αλλαγές, το κάνουμε ήδη και το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, τέτοιο τρόπο που δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν στην Ελλάδα. Ποτέ δεν είχαν ληφθεί τόσα πολλά μέτρα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Προφανώς το πρώτο το οποίο έπρεπε να κάνουμε είναι να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στην οικονομία μας και θα έλεγα την αξιοπιστία στη χώρα μας. Αυτό ήταν το άμεσο. Το μεσομακροπρόθεσμο είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές που θα μας φέρουν στην πορεία της ε, ανάπτυξης, ειδικά να αλλάξουμε το αναπτυξιακό μοντέλο. Εμεί ε, νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε μια οικονομία η οποία θα ανθίσει ειδικά όσον αφορά στην πράσινη οικονομία και στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της εκπαίδευση και τη υγεία, Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τεράστιο όλημα του υπερπολογισμού και αυτό απέτησε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσει που λαμβάνονται αυτή τη στιγμή και είναι πολύ σκληρές την περασμένη εβδομάδα πέρασαμε το πιο σκληρό πακέτο λιτότητας στην σύγχρονη ιστορία της ε, Ελλάδας και αυτό το κάνουμε όχι μόνο για να σώσουμε την οικονομία μας αλλά για να αποδείξουμε πως υπάρχει το απαραίτητο πολιτικό θάρρος και αξιοπιστία στη χώρα μας γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε τμήμα μια κοινότητας, της ευρωπαϊκής κοινότητας με την πραγματική έννοια του όρου, μια κοινότητα αξιών και θέλουμε και εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας μέσα σε αυτή την ευθύνη, που είναι, μέσα σε αυτή την κοινότητα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείχνουμε λοιπόν τη δέσμευσή μας για να προστατεύσουμε τη σταθερότητα του κοινού μα νομίσματος. Είπα στους Έλληνε ότι το 2010 θα πρέπει να είναι και θα είναι η χρονιά των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνηση, Αλλαγή του φορολογικού συστήματο, του συστήματο ασφάλεια. μείζονε αλλαγέ στη δημόσια διοίκηση, Μειώνουμε τα επίπεδα κυβέρνηση από τα 5 στα 3, αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα και φυσικά στο αναπτυξιακό μα μοντέλο. Αλλά όπω είπα, οι κοινωνικέ και θεσμικέ αλλαγέ δεν μπορούν να γίνουν τόσο γρήγορα όπως τα futures ή τα credit default swaps. Δεν μπορούμε αυτέ τι κοινωνικέ δεσμεύσει και τι πολιτικέ ευθύνε να τις, και τις συνήθειε και τα έθη να τα αλλάξουμε και του θεσμού που πρέπει να αλλάξουμε, να τα αλλάξουμε μία νυχτή. Χρειάζεται χρόνο για να το κάνουμε αυτό. Παίρνουμε άμεσα μέτρα, αλλά για να κάνουμε βαθύτερε διαρθρωτικέ και ουσιαστικέ αλλαγέ χρειαζόμαστε ε, χρόνο. Όχι πολύ χρόνο, αλλά χρειαζόμαστε χρόνο. Πιστεύω ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού υποστηρίζει αυτέ τι μεταρρυθμίσει. Είναι τολμηρέ μεταρρυθμίσει και φυσικά θα βοηθήσουν την οικονομία μα. Κάναμε αυτό που κάναμε. Αλλά αν εξακολουθήσουμε να δανειζόμαστε με υψηλά επιτόκια, και αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, δεν μπορούμε να μειώσουμε το χρέο μα. Ε, κάτι προσπαθούμε να κάνουμε αυτά σκληρά μέτρα. Στην πραγματικότητα, ζητάμε από το, το λαό μα, του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, να δεχθούν μειώσει μισθολογικέ για να μειώσουμε το έλλειμμα. Και αυτές οι θυσίες μπορούν να χαθούν πραγματικά σε μια στιγμή κερδοσκοπίας παγκόσμιες αγορές όπου κάποιοι πίσω από τους κομπιούτερ σε κάποια πόλη ίσως και εκτός της ε, Ευρώπης πιέζουν μερικά κουμπιά και όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε εμείς την ε, τσεπώνουν. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Δεν ζητάμε λοιπόν βοήθεια. Ο... Δεν είμαστε μία αήθης χώρα. Ε, μία χώρα που προσπαθεί να ζήσει από τον πλούτο των άλλων. Δεν ζητάμε χρήματα από τους Γερμανούς, τους Γάλλους ή τους Ιταλούς ή οποιουσδήποτε άλλου εργαζόμενου κάποιου άλλου λαού, από τους φορολογούμενους κάποιου άλλου λαού. Ζητάμε μια ισχυρή πολιτική στήριξη, ούτω ώστε να κάνουμε αυτές τι απαραίτητε μεταρρυθμίσεις και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα πληρώσουμε περισσότερο από το απαραίτητο, ούτω ώστε να ενεργοποιηθούν αυτέ οι μεταρρυθμίσει. Γι' αυτό λέμε, ας συνεργαστούμε, ας ανασκουμποθούμε ούτω ώστε να μην χρειαστεί να πληρώσουμε υψηλότερου φόρου, να μην έχουμε υψηλότερη ανεργία, να μην έχουμε πιο αργή οικονομική ανάκαμψη. Και αυτό συνέντε με το γεγονό ότι, όπω είπε και ο Υπουργό Οικονομικών πολύ σωστά, θα πρέπει ε, να αναγκάσουμε τις αγορές να ανταποκριθούν με θετικό τρόπο, έστω και πιεστικά. Η Ελλάδα είναι περίπου το 2% του κοινοτικού ΑΕΠ. Παρ' όλα αυτά, οι οικονομικές συνθήκες και η κατάσταση μπορεί να έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις από αυτό που υπονοεί αυτό το νούμερο, το 2%. Μπορεί να υπάρξει μια έτσι χιονοστιβάδα. Εμείς ε, έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε αυτή τη ρητορία, την καταστροφολογία, Παρ' όλα αυτά, αυτό το θέμα είναι ευρωπαϊκό. Η Ευρώπη χρειάζεται να πάρει δράση. Είμαστε και πολιτική ένωση και νομισματική ένωση. Και αυτό σημαίνει βαθύτερες σχέσεις και βαθύτερες και πιο ουσιαστικές αμοιβέ δεσμεύσεις για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα από κοινού. Έτσι, Στη συζήτηση που γίνεται ανά τον κόσμο για το αν η Ευρώπη θα αποτύχει, αν θα σβηστεί από το χάρτη, εγώ θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Γιατί, καταρχά, παρότι η Ευρώπη είναι ένα τεράστιο στοίχημα, ένα φιλόδοξο στοίχημα, στην πραγματικότητα στο μυαλό μου είναι ένας πρόδρομος του γιατί χρειαζόμαστε μια ευρύτερη παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Είμαστε μια ένωση 27 κρατών, 16 είμαστε στην Ομοιοσματική Ένωση, έχουμε ο καθένας τη γλώσσα μας, τις εμπειρίες μας, ο καθένας έχουμε την ιδιοσυγκρασία του. Αλλά έχουμε σφραγίσει τις μοίρε μας μέσα στον ίδιο κύκλο. Και από κοινού προσπαθούμε, ε, παραχωρώντας ένα τμήμα της κυριαρχίας, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Ε, μετά το Παγκόσμιο Πόλεμο η Ευρώπη είναι ένας καταλήτης για να εμβαθύνουμε τις διαδικασίες ε, ολοκλήρωσης και να βρούμε λύσεις. Το θέμα είναι και πώς θα βρούμε λύσεις και πώς θα αντιμετωπίσουμε την παγκοσμιοποίηση γενικότερα σε πιο παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Θα ήθελα να ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας ο, αυτό που είπε ο Ντομινίκ Στροσκάν χθες. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία να ρυθμίσουμε το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εμείς στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας και τα αντιμετωπίζουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο ad hoc, όπως προκύπτουν. Αλλά αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε για, τα για το είδος των φορέων και θεσμών που χρειαζόμαστε, ε, ίσως ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Γίνεται λόγος γι' αυτό Ποιο θα είναι το περιεχόμενό του, πώς θα δουλέψει. Αυτό είναι ένα θέμα προσυζήτηση. Είναι τεράστια αυτά τα θέματα, πολύ σημαντικά. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να μπουν επιτάπητος αν θέλουμε να εμβαθύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνεργασία μα. Όμω αυτά είναι θέματα τα οποία δεν αντιμετωπίζουν τα άμεσα προβλήματα τα οποία έχουμε. Αυτά τα αντιμετωπίζουμε παίρνοντα τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε. Παράλληλα, όμω, θα πρέπει να μπορούμε να δανειζόμαστε με φυσιολογικά επιτόκια ανάλογα με αυτά που οι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε και οι χώρε τη Νομισματική Ένωση ε, δανείζονται. Σα ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα. Σα εύχομαι επιτυχία στο δύσκολο καθήκον σα, στο δύσκολο έργο σα και είμαι έτοιμο να ακούσω όχι μόνο τι ερωτήσει σα, αλλά και τι υποδείξει σα. Γιατί εδώ είμαστε μια οικογένεια, μια ένωση και προσπαθούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύσκολα προβλήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ και για την ευκαιρία που δίνεται στους συναδέλφους να κάνουν ερωτήσεις. Θα θέλαμε εμείς ε, όλες οι πολιτικές ομάδες να μπορέσουν να κάνουν ερωτήσεις, οπότε θα δώσω τον λόγο σε κάθε ομάδα και στον ε, βουλευτή που έχει πει πως θέλει να κάνει ερωτήσεις. Να τονίσω ένα πράγμα, συνάδελφοι. Ο χρόνος πιέζει, οπότε παρακαλώ να περιοριστείτε στο ένα λεπτό. Ξεκινάω με τον κύριο Σκυλακάκη από το ΕΛΚ. Καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Από τη δημιουργία της Ευρωζώνης μέχρι σήμερα έχει σχηματιστεί ένα χάσμα ανταγωνιστικότητας, κυρίως μεταξύ της Γερμανίας και μια σειράς χωρών του Νότου. Ένα μέρος της λύσης θα μπορούσε να ήταν η αύξηση των μισθών και της κατανάλωσης στη Γερμανία. Ένα άλλο μέρος διαρθρωτικές αλλαγές στις χώρες που έμειναν πίσω στην ανταγωνιστικότητα. Από τη δική σας πλευρά, από την ελληνική πλευρά, τι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σκέπτεστε να πάρετε για να βελτιώσετε την ελληνική ανταγωνιστικότητα και να συνεισφέρετε σε αυτή την προσπάθεια. Και μία δεύτερη πτυχή σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθεί στο μέλλον. Θέλουμε ένα πιο χαλαρό σύμφωνο σταθερότητας το, ή ένα σύμφωνο σταθερότητας που θα εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ποδηματά. Ε, Πρόεδρε, Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα την ε, πολιτική μας ομάδα και ιδιαίτερα τον ε, συντονιστή μας, τον Σέντζο Κονφεράτη, που με όρισε ε, ως μία εκ των ομιλητών στην απόψινή ακρόαση. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση που αντικατοπτρίζει τις απόψεις της πολιτικής μας ομάδας συνολικά. Η ομάδα λοιπόν των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχει υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή της κρίσης, κύριε Πρόεδρε, την ανάγκη συγκρότησης στο ευρωπαϊκό επίπεδο ενός μηχανισμού υποστήριξης των χωρών μελών με μεγάλες δημοσιονομικές δυσκολίες αλλά και σταθεροποίησης του ευρώ. Ο πρόεδρος, ε, ο Ράσμουσεν μαζί με την Περβάνς Περές έχουν αρθρογραφήσει σχετικά στον ευρωπαϊκό τύπο. Κάποιοι άλλοι όμως εταίροι υποστηρίζουν ότι εκείνο που μας λείπει δεν είναι ένας μηχανισμός αλληλεγγύης και υποστήριξης αλλά ένας μηχανισμός ακόμα περισσότερο αυστηρής επιτήρησης και τιμωρίας που θα φτάνει μέχρι και την έξοδο από τη ζώνη του ευρώ για χώρες με παρατεταμένη δημοσιονομική εκτροπή. Εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν είναι αν θεωρείτε ότι αυτές οι εκδιαμέτρου διαμέτρου διαφορετικές απόψεις αντικατοπτρίζουν και αντανακλούν τελικά ριζικά διαφορετικές αντιλήψεις για το παρόν και το μέλλον της ζώνης του ευρώ. Σας ευχαριστώ πολύ. χωρίς μικρόφωνο. Είπα να μιλήσω και μια γλώσσα την οποία ξέρετε και εσείς ε, κύριε Πρωθυπουργέ, τα σου ειδικά. Σας ε, καλωσορίζω λοιπόν. Εσείς ε, είστε τίμιος. Έχετε όλοι μας την υποστήριξη και η Σουηδία χρειάστηκε κάποτε να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση. Ξέρουμε τι σας περιμένει και παρακολουθούμε από πολύ κοντά τη δουλειά σας. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα πλήττει κυρίως την Ευρωζώνη αλλά και τις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Ε, εγώ και ο και εσείς κύριε Πρωθυπουργέ είμαστε από τους ε, μεγάλους υποστηρικτές ε, του ευρώ έστω ε, και αν η χώρα μου βέβαια δεν είναι στην ευρωζώνη. Τι σημαίνει η κρίση της Ελλάδας για τις χώρες εκτός ευρωζώνης θα είναι ένα κίνητρο για να μην γίνουν μέλη της ευρωζώνης. Λοιπόν, εσείς θεωρείτε κύριε Πρωθυπουργέ ότι η κρίση στην Ελλάδα οφείλεται στο ότι το ευρώ είναι νόμισμα και θα θέλατε να μην είχε μπει ποτέ η Ελλάδα στην ευρωζώνη. Ε, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας, ε, βεβαίως ε, τα θέματα τα οποία ακούει κανείς συνήθως είναι ότι έχουμε μια αύξηση μισθών ιδιαίτερα στο δημόσιο τα τελευταία χρόνια ως ένα βασικό στοιχείο της μείωσης της ανταγωνιστικότητας εγώ θα έθετα όμως ε, το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας σε άλλους τομείς. Εγώ νομίζω ότι ε, θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει μια ε, ιδιαιτερότητα ότι έχουμε πράγματι έναν πολύ μεγάλο, χαλαρό και, και, και δαπανηρό δημόσιο τομέα αλλά λόγω της, της μεγάλης γραφειοκρατίας και πίσω από τη γραφειοκρατία πολλές φορές ακόμα και, προβλήματα ε, διαφθοράς. Αυτό όμως μας δίνει και τα απαραίτητα περιθώρια να κάνουμε σοβαρές ε, μειώσεις με διαρθρωτικές αλλαγές, μειώσεις στη γραφειοκρατία, μειώσεις με την απλοποίηση των διαδικασιών, όπως τώρα πάμε σε ένα φορολογικό σύστημα πιο απλό, όπως πάμε σε ένα σύστημα διοικητικό πολύ πιο απλό, κόβοντας από πέντε επίπεδα της, ε, της διακυβέρνησης της χώρας μας σε τρία, δηλαδή στο κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό, ε, συνενώνοντας πολλούς δήμους, καταργώντας πολλές ε, εταιρείες δημοτικές, επιχειρήσεις δημοτικές, αλλά και συγχωνεύοντας πολλές υπηρεσίες κεντρικές που δεν έχουν λόγο ύπαρξης κάνοντας οικονομίες ε, ε, με τη διαφάνεια. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, στον χώρο των νοσοκομείων τεράστια προβλήματα κόστους λόγω ε, της αδιαφάνειας, της διαχείρισης και δυστυχώς μιας συνενοχής μεταξύ ενός μεγάλου μέρους του ιατρικού προσωπικού και των φαρμακευτικών βιομηχανιών όπου ακόμα και ο ΩΣΑ μας λέει με μελέτες ότι θα μπορούσαμε να μειώσουμε το κόστος της δαπάνης της και να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα κατά 30 με 50% και αν σκεφτείτε ότι ε, σήμερα έχουμε ένα χρέος στο νοσοκομεία κοντά στα 7 δισεκατομμύρια, αυτό θα ήταν, αυτή η μείωση θα ήταν το μισό τουλάχιστον από αυτό το οποίο εξοικονομήσαμε με, την μείωση, με, τα, με αυστηρά μέτρα τα οποία έχουμε πάρει αυτή την, αυτή την εποχή. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η βοήθεια στην η ανταγωνιστικότητα από τη μια μεριά θα είναι σημαντική, ε, ε, ο σημαντικός εξυγχρονισμός του δημόσιου τομέα. Δεύτερον, ε, η βοήθεια στην, στην ανάπτυξη νέων τομέων ή στην καλυτέρευση, στην βελτίωση τομέων όπως είναι του τουρισμού, που είναι ένας δυναμικός τομέας, πηγαίνοντας προς την πράσινη ανάπτυξη με νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση, αλλά και στην υποστήριξη νέων επιχειρήσεων με την βελτίωση Σβήστε το μικρόφωνο του κύριου Παπανδρέου. Uh, I'll, I'll continue in English. Uh, on, on the issue of the, uh... Για το θέμα της συνθήκης του Μάστριχτ και αν είναι πολύ αυστηρή ή πολύ ελαστική. Πρέπει να εξετάσουμε τους διάφορους θεσμούς που δεν υπάρχουν σε αυτό το σημαντικό στίχημα που είναι το ευρώ και η ευρωζώνη. Καταρχάς, πέρυσι, μετά την κρίση, υπήρξε μια χαλαρότητα που ονομάστηκε ευελιξία για τα κριτήρια του Μάστρικτ. Εγώ ήμουν στην αντιπολίτευση τότε. Και είχα συναντηθεί με τον Χωσέ Μανουέλ Μπαρόζο και του είπα δεν μου αρέσει η λέξη ευελιξία. Μπορεί να φαίνεται περίεργο από το στόμα ενός σοσιαλιστή, αλλά τι εννοούσε στην πραγματικότητα. Ότι αν έχουμε λύματα υψηλότερα από αυτά που επιτρέπουν τα κριτήρια του Μάστερ, κανένα πρόβλημα. Ούτω ή άλλω όλε οι χώρε, όλε οι αναπτυγμένε χώρε και ακόμη και αναπτυσσόμενε χώρε, και αναδυόμενε οικονομίε το ίδιο κάνανε. Λέγανε ότι θα πρέπει να βάλουμε χρήμα στην οικονομία μα, να ρίξουμε χρήμα στην οικονομία μα, θα πρέπει Βεβαίω με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε κάποια ελλείμματα, αλλά δεν θα μπούμε σε ύφεση. Θα τονώσουμε την οικονομία μα. Ε, αυτό έγινε και στι ΗΠΑ, έγινε και στην Ευρώπη. Είπα λοιπόν, α είμαστε συγκεκριμένοι, α πούμε ότι όλοι θα έχουμε μία αύξηση 3% ή 4% ή 2% ό,τι συμφωνήσουμε. Να το κάνουμε συντονισμένα και υπό την εποπτεία της Κομισιόν για να δούμε πού πάνε αυτά τα χρήματα. Αν πούμε απλώς ευελιξία, τότε θα δώσουμε ένα μήνυμα, ένα σήμα σε κάποιες χώρες και αυτό το μήνυμα μπορεί να σημαίνει τελικά ότι θα αυξηθούν ανεξέλεγκτα τα ελλείμματα, γιατί αυτό συνέβη στην Ελλάδα τελικά. Χρειαζόμαστε περισσότερο ε, συντονισμό και βεβαίως χρειαζόμαστε ευελιξία λόγω της κρίσης, αλλά όλα αυτά, ε, όλη την προσπάθεια να την κάνουμε πιο οργανωμένα, πιο συντονισμένα η ιδέα ενός μηχανισμού υποστήριξης είτε ονομάζεται ε, Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο είτε οτιδήποτε άλλο είναι πολύ σημαντικό. Η κυρία Μπερές και άλλοι το ανέφεραν ότι είναι σημαντικές ιδέες. Υπάρχουν και άλλες ιδέες που, που κυκλοφορούν και συζητιούνται. Αλλά αυτά όλα θα πρέπει να γίνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Φυσικά κάποιο μπορεί να τιμωρηθεί με βάση τα κριτήρια του Μάστρικ λόγω τη κακή του διαγωγής. Και μάλιστα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που μπορούν να προσδιορίζουν σε τι θα συνίστανται αυτές οι τιμωρίε. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και οι χώρε που έχουν προβλήματα και που κάνουν προσπάθεια για να τα επιλύσουν υποστηρίζονται για να εφαρμοστούν τα προγράμματά του και να είναι αποτελεσματικά. Γιατί το να τιμωρούμε απλώς, ίσως δεν είναι η λύση. Και τελικά η τιμωρία και η αποπομπή θα είναι αποτυχία, όχι μόνο για τη χώρα αυτή, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, να πω στο Σουηδό φίλο και το θέμα που έθεσε για την Ευρωζώνη. Για την Ελλάδα, η Ευρωζώνη ήταν κάτι το θετικό. Καταρχάς, σταθεροποίησε το νόμισμά μας, γιατί το νόμισμά μας έγινε το ευρώ και δεύτερον μας βοήθησε να αναπτυχθούμε Τα πρώτα χρόνια του ευρώ είχαμε σημειώσει μια σημαντική ανάπτυξη. Και σήμερα ακόμα είναι σημαντικό. Βεβαίως, και αυτό είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, υπάρχει η έλλειψη ενός μηχανισμού. Αν δεν είμαστε, ας πούμε, στην ε, Ευρωζώνη, σήμερα α, αυτά τα μέτρα που πήραμε μας θα μας τα είχε ζητήσει και το Διεθνές Συμπισματικό Ταμείο να τα, να τα πάρουν. Και η Κομισιόν τις τελευταίες ε, εβδομάδες ε, παρακολουθούσε τη χώρα μας μαζί με την Κεντρική Τράπεζα, συμφώνησε με αυτά τα μέτρα και το IMF συμφώνησε με αυτά τα μέτρα. Ε, ουσιαστικά είμαστε στα πλαίσια ας πούμε, επιτήρησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, παρότι δεν το λέμε έτσι. Απ' την άλλη δεν έχουμε τις διευκολύνσεις που δίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα χρήματα, παραδείγματο χάρη, αν τα χρειαστούμε. Εμεί λέμε ότι δεν τα χρειαζόμαστε, αλλά αν τα χρειαστούμε δεν τα έχουμε. Και επίση έχουμε ένα περιορισμό που άλλε χώρε, ε, γιατί ήμουνα στην Ουγγαρία πριν από δύο μέρε, η οποία δεν είναι στην Ευρωζώνη και έχει τη δυνατότητα να παίξει με το νομισμά τη. Αυτό είναι ένα διορθωτικό μηχανισμός όταν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν λοιπόν δύο θέσμες μέτρων. Εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε να μπούμε σε μια κατάσταση όπου έχουμε τις τιμωρίες που προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά καθόλου τα πλεονεκτήματα της Ευρωζώνης. Εδώ θα πρέπει να παίξει το ρόλο της Ευρωπαϊκή Ένωση και να πει μπορούμε εμείς να υποκαταστήσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, έστω και ad hoc ή αλλιώς η Ελλάδα θα πρέπει να έχει την επιλογή να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ελπίζουμε βεβαίως να, μην κατασ... να μην χρειαστεί κάτι τέτοιο. Περνάμε στον επόμενο γύρο των ομιλητών. Παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο, Πασκαλ Καρφά. Και μετά ο κύριος Χουντής Καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ, εξ ονόματος της ομάδας ε, των Πρασίνων ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας ε, στις εργασίες Επιτροπής μας. Θέλω να επανέλθω στο Σύμφωνο Σταθερότητας και στα διδάγματα που θα πρέπει να ανασύρουμε από την ελληνική κρίση και την κρίση γενικότερα. Ένα από τα προβλήματα της Ευρωζώνης είναι ότι μετά από τη δημιουργία του ευρώ το έλλειμμα ορισμένων χωρών αυξήθηκε ενώ τα πλεονάσματα του ισοζυγίου, του τρέχοντος ισοζυγίου των άλλων χωρών, άλλων χωρών της Ένωσης αυξήθηκαν σημαντικά. Λοιπόν, υπάρχει μια ανισορροπία. Δεν φαίνεται από την κρίση ότι τελικά το σύμφωνο σταθερότητας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα νέο κριτήριο καταμερισμένης διαχείρισης και παρακολούθησης του ισοζυγίου τρεχουσών πληρωμών τόσο για τα πλεονάσματα όσο και για το ελλείμματα. Ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να σας καλωσορίσω εκ μέρους της Ενωτικής Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να σας ευχαριστήσω για την ομιλία και να υπογραμμίσω το γεγονός ότι διαλέξατε αυτή την Επιτροπή που ασχολείται με την κρίση για να συζητήσετε μαζί μας. Η ερώτησή μου είναι, υπάρχει σαφές και συγκεκριμένο σχέδιο στήριξης της ελληνικής οικονομίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι μέχρι τώρα στάση και οι δηλώσεις των ηγετών μάλλον ενισχύουν την κερδοσκοπία. Αν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, τίθενται όροι παρόμοιοι με τους όρους που θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε πιθανή προσφυγή σε αυτό, δηλαδή σκληρότερα μέτρα σε βάρος των εργαζομένων από αυτά που έχετε ήδη λάβει και σε μια τέτοια περίπτωση κύριε πρωθυπουργέ πιστεύετε ότι με τέτοια μέτρα μπορεί να αντιμετωπιστεί η ύφεση μπορεί να αντιμετωπιστεί η απασχόληση. τέλος θα διεκδικήσετε μια άλλη νομισματική πολιτική που να εξασφαλίζει μηχανισμό δανεισμού τελευταίας καταφυγή και θα αντιμετωπίζει την κερδοσκοπία. ευχαριστώ πολύ. ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ. Εσείς ε, δεν υποστηρίζετε ότι τελικά αυτά τα δρακόντια μέτρα τα οποία αναλαμβάνετε ε, αντί να λύσουν τα προβλήματα θα πνίξουν ακόμη περισσότερο την Ελλάδα που όλοι μας ε, θέλουμε να προστατεύσουμε. Η Ελλάδα μήπως χρειάζεται καλύτερα ένα, μια, μια συγκράτηση της δαπάνης ως ε, λύση και αντί αυτής της μείωσης της δημόσιας δαπάνης ε, δεν θα έπρεπε να λάβουμε άλλα μέτρα όπως είναι η πρόθεση του τουρισμού ας πούμε όπως ε, με δημιουργία επίσης ενός εθνικού νομίσματος το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί παράλληλα εσωτερικά χωρίς να βγείτε από το ευρώ και αυτό βάσει του, ε, άρθρου 50 της συνθήκης χωρίς ε, αυτήν την, πολιτική της πραγματικής νομισματικής προστασίας μπορείτε να φανταστείτε ένα άλλο μέλλον για την Ελλάδα που να μην μοιάζει με εκείνο Υπάρχει κι άλλος ένας γύρος από τρεις ομιλητές. Μπορείτε να απαντήσετε τώρα. Για το θέμα του ελλείμματος των τρεχουσών πληρωμών. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταστήσουμε την οικονομία, την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική. Φυσικά ε, υπάρχει και το θέμα τη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία. Αλλά υπάρχουν ανισορροπίε και σε, όλο τον κόσμο. Σε νομίσματα, ορισμένα θεωρούνται υποτιμημένα και θα πρέπει να τιμηθούν. και με τις αλλαγές μπορεί να δημιουργήσουν ε, τεράστια προβλήματα για, για την ανταγωνιστικότητα. Αλλά με τη ζήτηση μπορεί να δημιουργηθεί, να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ανάπτυξη στον πλανήτη. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, έχουμε την ευθύνη να κάνουμε τις απαραίτητες ε, μεταρρυθμίσεις για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Ο κ. Χουντής είπε ότι αυτά τα μέτρα που πήραμε δεν είναι μέτρα τα οποία από μόνα τους θα μας βγάλουν από την κρίση και θα μας βάλουν σε, μια τροχιά ανάπτυξης. Ε, η συνθήκη του Μάστριχτ λέει σταθερότητα και ανάπτυξη και τα δύο. Η ανάπτυξη είναι η άλλη όψη του νομίσματο. Και εδώ χρειαζόμαστε να κάνουμε τι απαραίτητε επενδύσει, Θα επενδύσουμε από τα διαφορετικά ταμεία και το Ταμείο συνοχή. Υπάρχουν χρήματα που θα επενδυθούν σε υποδομές και κατάρτιση για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Επίσης πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει μεγάλο δυναμικό για να γίνει μια πράσινη οικονομία. Έχουμε το υψηλότερο δυναμικό στην Ευρώπη σε ολική ενέργεια, αλλά δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει. Δεν έχουμε επενδύσει αυτό το δυναμικό τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι κάποιοι τομεί όπου μπορούμε να στραφούμε και να επενδύσουμε. Επίσης, ε, έχουμε λάβει μέτρα επίπεδου διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Ε, μιλήσαμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν θα ζητούσαν κάτι παραπάνω. Αν πάμε σε αυτού, δεν θα μα δείσουν κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη κάναμε. Αλλά εγώ θα προτιμούσα μια ευρωπαϊκή λύση. Θα προτιμούσα μια ευρωπαϊκή λύση ω ε, μια και είμαστε τμήμα τη Ευρωζώνη, επειδή είμαι λαύρο ε, ευρώφιλο και ευρωπαίο και γιατί θέλω να δείξω στον κόσμο ότι η Ευρώπη μπορεί να δράσει μαζί, συντονισμένα. Δεν ζητάω χρήματα, όπως είπα. Αλλά θέλουμε πάνω στο τραπέζι ένα κάποιο εργαλείο ένα μέσο. Και αυτό το δάνειο νομίζω ότι θα αρκέσει για να εξασφαλίσει ότι τα spreads και οι κερδοσκόποι θα φύγουν, θα μας αφήσουν ήσυχου. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κερδοσκοπίας απέναντι στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα ευρύτερο θέμα. Γι' αυτό λέω, ας χρησιμοποιήσουμε την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να να αντιμετωπίσουμε τελικά τα βαθύτερα προβλήματα που υπάρχουν παντού και στην Ευρώπη και θα τα αντιμετωπίσουμε πολύ πιο έντονα στο μέλλον. Για την υποτίμηση και την δημιουργία ενό εθνικού νομίσματο τελικά. Νομίζω ότι παίρνουμε, έχουμε πάρει ήδη τα απαραίτητα μέτρα, ούτω ώστε η οικονομία μα να μπει σε μια τάξη και να αντιμετωπίσουμε τα, τα θέματα μέσα στο πλαίσιο της συνθήκης του Μάστριχ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πάρουμε άλλα μέτρα. Και θα ήταν πάρα πολύ περίπλοκο να μπούμε τώρα σε μια κατάσταση με ευρώ και ένα εθνικό νομίσμα παράλληλα. Νομίζω θα στέλναμε και ένα λάθος μήνυμα για το και το μέγεθος των προβλημάτων που έχουμε. Έχουμε προβλήματα, αλλά δεν πρόκειται να χρεοκοπήσουμε. Θα επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα και έχουμε ένα τεράστιο δυναμικό ως οικονομία και υπάρχουν τομείς ανάπτυξης. Ας μην φτιάξουμε μία εικόνα ότι είμαστε στο χείλος Σαββίσου. Γιατί έχουμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα και νομίζω ότι θα προχωρήσουμε. Uh, Γυρνάει ο τελευταίο κύκλο ερωτήσεων. Χάνς Πέτερ Μάρτιν, Ότ Μαρκάρα και Περβάνο Περέ. Ναι. Εγώ είμαι υπερασπιστής ε, του ευρώ και φιλοευρωπαίος αυστριακός, αλλά γι' αυτό ακριβώς, κύριε Πρόεδρε, είμαι επικριτικός, γιατί σωστά είπατε ότι δεν υπάρχει αρκετός έλεγχος. Θα ήθελα Ακριβώς από αυτή τη βάση των διαφόρων που ακούστηκαν να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Αντιληφθήκαμε πως ε, η συζήτηση που γίνεται στη Γερμανία μεταφέρθηκε στην Ελλάδα, όμως αυτό το οποίο διάβασα από σας είναι πως από ό,τι φαίνεται δεν τελειώνει. Πρώτα απ' όλα, θεωρείτε πως η συζήτηση αυτή έχει ε, τελειώσει όσον αφορά τυχόν εγγύηση από Γερμανίας. Ερώτηση δεύτερη θεωρείτε πως θα ήταν ε, σωστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να κάνουμε μια εξεταστική των, των πραγμάτων επιτροπή για να δούμε ποια είναι τα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από την Ελλάδα και για πιθανές άλλες περιπτώσεις όπως παραδείγματος χάρη την Ισπανία. Και τρίτον, θέσαμε ερωτήματα προς την ε, Κομισιόν και προέκυψε πως υπήρξαν Κάποιε ε, παρατυπίες στην Ελλάδα 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και ο Όλαφ, η υπηρεσία καταπολέμησης απάτη δεν έχει μπορέσει να ανακτήσει ούτε το 1 τρίτο ακόμα. Τι θα κάνετε σχετικά με αυτό. Ότμαρ Κάρα, κύριε Πρωθυπουργέ, πρώτα απ' όλα σας ε, καλωσορίζω και εξ του ΕΛΚ να σας πω πως ε, θεωρώ την δουλειά σας ε, εξαιρετική και τι δηλώσει σας ε, σαφέστατε και μπορούμε να σα διαβεβαιώσουμε πως η Ελλάδα είναι μέλος της ε, κοινότητάς μας και βεβαίως γνωρίζουμε την ευθύνη που έχουμε για μια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχουμε τρία επίπεδα. Ελλάδα, Ευρώπη και τους παγκόσμιους κανόνες. Από αυτά τα οποία μας είπατε σήμερα αντιλαμβάνομαι πως είστε ικανός και θέλετε να κάνετε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και θεωρείτε πως μπορείτε να τα καταφέρετε μόνοι σας. Το δεύτερο είναι πως αντλείτε τα διδάγματα που πρέπει για το τι πρέπει να γίνει και τι λείπει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να βοηθούμε σε τέτοιες κρίσεις και να μην καταφύγουμε σε τυχόν άλλε ευρύτερε λύσει στο παγκόσμιο επίπεδο. Και τρίτον, χρειαζόμαστε παγκόσμιου κανόνε. Οπότε θέλω από εσά να γνωρίζω τι δεν μπορείτε να λύσετε μόνοι σα επιτόπου στην Ελλάδα με του κανόνε που έχουμε και πού πρέπει βραχυπρόθεσμα να φανούμε αλληλεγγύοι. Κύριε Περβάνσο. Κύριε Πρωθυπουργέ, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε από μόνο σας ότι τα θαραλέα μέτρα τα οποία έχετε αναλάβει προκαλούν το θαυμασμό μας. Η κρίση πολλές φορές μπορεί να δημιουργεί νέες ευκαιρίες αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να οδηγεί και σε βιαστική λήψη μέτρων που μπορεί να είναι αντιπαραγωγικά. Λέτε εσείς ότι η χώρα σας είναι υπεύθυνη λόγω της έλλειψης εσωτερικών διαρθρωτικών αλλαγών. Μα και η χώρα μου όμως είναι υπεύθυνη για το δημόσιο χρέος της. Διότι όπως είπε και κάποιος κυβερνητικός εκπρόσωπος χοροπηδούσε ως κατσίκι χωρίς ποτέ να παίρνει στα σοβαρά το έλλειμμα και το σύμφωνο σταθερότητας. Η Ελλάδα δράτει αυτή την ευκαιρία σήμερα και συμμερίζομαι εγώ την άποψή σας. Λοιπόν υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ. Το ελληνικό ζήτημα από τη μια και η Ευρωζώνη θα υποστηρίξει με όλες τις, τις δυνάμεις τα θαραλέα μέτρα που αναλαμβάνεται. Και σε μια δεύτερη φάση η ήρεμα να προβληματιστούμε για το τι συνέβη αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια όπου οι διαφορές μεταξύ των οικονομιών οξύνθηκαν στην ευρωζώνη και έγινε η έκρηξη της ελληνικής υπόθεσης. Τελικά ρωτώ πότε λέτε εσείς να ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη φάση κύριε Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ. για τις αποζημιώσεις. Είναι ανοιχτό θέμα. Ε, κατά καιρούς το έχουμε συζητήσει με τη Γερμανία. Ότι, νομίζω όμως ότι σε αυτή τη φάση είναι άκερο να το θέσω επιτάπητος. Συζητάμε για άλλα θέματα. Θα περιπλακούν τα πράγματα. Και θα δώσω και ένα μήνυμα ότι δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε στη χώρα. Να προβούμε στις αλλαγές. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν ψάχνουμε από διπομπέους τράγους. Δεν ψάχνουμε τρόπους και λόγους να αποφύγουμε τα επώδυνα μέτρα. Τα προωθούμε. Είναι τα πιο δύσκολα μέτρα που έχει λάβει ποτέ η Ελλάδα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Και επομένως, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι και το στέλνουμε και δεν δεν είναι δικό μου κουράγιο αυτό. Είναι το κουράγιο του ελληνικού λαού που το καθιστά δυνατό. Ότι δηλαδή μπορούμε να τακτοποιήσουμε τα της Ελλάδας, τα του οίκου μας. Έπειτα, εμείς οι ίδιοι έχουμε ξεκινήσει μια εκταστική επιτροπή για αυτό το θέμα. Υπάρχει μια εξεταστική επιτροπή στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις πρακτικές των τραπεζών για την Ελλάδα, παρότι οι πρακτικές θεωρούνταν πολύ αξιόπιστες και η Ελλάδα χρησιμοποίησε πρακτικές που δεν ήταν κρυφές. Φυσικά οι τράπεζες οι οποίες επέστρεψαν στα συνήθη δεν ήταν οι καλύτερες. Ε, οι πρακτικές αυτές δεν ήταν οι καλύτερες. Γιατί οδήγησαν στην κρίση. Και θέλω να τονίσω κάτι τώρα εδώ. Ότι η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωζώνη χωρίς μαγειρέματα με την αξία της, με το σπαθί της. Παρότι άλλαξε τα λογιστικά για τους εξοπλισμούς, υπάρχουν δύο τρόποι για να αποτιμήσεις ε, τη σημασία των εξοπλισμών. Είτε τους βάζεις στον προϋπολογισμό, είτε Δηλαδή, του βάζει στον προπολογισμό όταν παίρνει τα όπλα και ο άλλος τρόπος, όταν δίνεις την παραγγελία. Εμείς το κάναμε όταν πήραμε τα όπλα. Τώρα θα κάνουμε το αντίθετο. Όταν, θα το κάνουμε όταν δώσουμε την παραγγελία. Η προηγούμενη κυβέρνηση άλλαξε τα πράγματα. Όταν παίρνεις τα όπλα, δεν χρησιμοποιούμε την πρακτική της καταχώρησης όταν παίρνει τα όπλα, αλλά όταν περνά την παραγγελία. Όταν δίνεις την παραγγελία. Αυτό τι σημαίνει. Ότι η Ελλάδα όταν μπήκε στην Ευρωζώνη μπήκε με ένα έλλειμμα 3,1. Είμαστε πολύ κοντά στο 3%. Άλλες χώρες είχαν μπει με 3,3, 3,5 Υπάρχει λοιπόν ένας μύθος ότι η Ελλάδα τότε δεν ήταν εντάξει. Φυσικά όταν έχει τόσο μεγάλο στοτιωτικό προπολογισμό και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε. Θέλουμε να το μειώσουμε αυτόν τον προπολογισμό και ελπίζουμε μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό ειρηνευτικό σχέδιο να εξομαλύνουμε και τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Και τότε αυτό θα είναι η μεγαλύτερη βοήθεια για τον ελληνικό προϋπολογισμό. Έχουμε ένα προπολογισμό όπου το 4-5% του ΑΕΠ πηγαίνει στου εξοπλισμού. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό στην Ευρωζώνη ή στην Ευρώπη. Μην το ξεχνάμε λοιπόν αυτό. Για το θέμα της αλληλεγγύης. Ευχαριστώ κύριε Καράς. Έχετε δίκιο. Κάναμε τη δική μας την προσπάθεια. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να πολεμήσουμε τις δυνάμεις της αγοράς, ειδικά αν κερδοσκοπούν. Και εκεί χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Ίσως η ελληνική περίπτωση είναι εξαιρετική, αλλά δεν είναι η μόνη εξαίρεση. Ίσως είναι ακραία, αλλά δυστυχώς έχουμε δει κι άλλες τέτοιες πρακτικές ανά τον κόσμο. Υπάρχει πολύ κερδοσκοπία. Μετά την κρίση χρειαζόμαστε να ρυθμίσουμε τις αγορές, λοιπόν. Πρέπει να τις ρυθμίσουμε. Ορισμένοι λένε ότι δεν πρέπει να έχουμε κανόνες. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να πιέσουμε τους αγορές που να ασφικτιούν. απλώ να τις ρυθμίσουμε. Δεν μας αρέσουν ε, τα φανάρια, γιατί μειώνουν ταχύτητα των αυτοκινήτων, αλλά εμποδίζουν και τα ατυχήματα. Ε, γι' αυτό λοιπόν δεν θέλουμε και στα χρηματοπιστωτικά ε, ατυχήματα όπως η κερδοσκοπία. Τέλο πάντων, πιστεύω ότι αυτή η κρίση και για την Ελλάδα είναι μια ευκαιρία. Είναι μια δύσκολη, επώδυνη κρίση, αλλά θα την χρησιμοποιήσουμε ως ευκαιρία για ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα, για μια καλύτερη, πιο ανταγωνιστική οικονομία, για μια οικονομία η οποία θα μας κάνει περήφανους. Και εμάς τους Έλληνες και εσάς τους Ευρωπαίους. Και αυτή η θέληση υπάρχει στην Ελλάδα. Παρότι αυτά τα μέτρα είναι επώδυνα, ο κόσμο λέει ναι, χρειαζόμαστε αυτή την αλλαγή. Σε οποιονδήποτε και να μιλήσετε, αυτό θα σα πει. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία παρά την επώδυνη. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, α χρησιμοποιήσουμε αυτή την συγκυρία ευκαιρία. Χάρηκα που ήρθα εδώ σήμερα. Σας εύχομαι πραγματικά καλή τύχη για να βρούμε τις καλύτερες λύσεις. Ελπίζω αυτή η Επιτροπή να παίξει τον κρίσιμο ρόλο της αυτή την ιστορική στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για να δούμε τι πολιτικές θα προχωρήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τη χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά και τις κοινωνικές πολιτικές μαζί με τις οικονομικές. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε κύριε Πρωθυπουργέ πόσο εκτιμήθηκε η παρέμβασή σας. Προτείνω διάλειμμα 5 λεπτών να συνοδεύσει τον κύριο Πρωθυπουργό στην πόρτα.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 Λοιπόν, όσοι δεν θέλουν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση, παρακαλώ να φύγουν σιγά σιγά και να μην συζητάνε τουλάχιστον μέσα στην αίθουσα. Uh, Έχουμε τώρα το πρώτο πάνελ ε, της ημέρας με τίτλο «Σύμφωνο σταθερότητας ανάπτυξης και μεταρρύθμιση και βιωσιμότητα των δημοσίων δαπανών». Έχουμε τρεις ε, εξέχοντες ομιλητές, τα βιογραφικά του σημειώματα τα έχετε, οπότε δεν πρόκειται να σας πω το τι κάνουμε. Έχουμε στα αριστερά μας τον κύριο Λουκα Τσούκαλη, καθηγητή στο Καποδιστριακό, κατόπιν ο Ζαν Πιζανή, ε, καθηγητής στο Παρίσι και Μπρόγγελ και μετά την κυρία Ντανιέλα Σβάρτσερ από το Βερολίνο, επικεφαλής της ερευνητική μονάδας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ολοκλήρωση. Έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είναι τιμή μου που με καλέσει να απευθυνθώ στα μέλη της Επιτροπής σας και στον χρόνο που μου αναλογεί θα κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις για τις συνέπειες της κρίσης για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και την διακυβέρνηση της, Ευρωπαϊ... της Ευρωζώνης συγκεκριμένα. Η αφετηρία μου είναι ότι αυτό το οποίο ξεκίνησε ως δημοσιονομική κρίση εξαπλώθηκε στην πραγματική οικονομία και αποτελεί το τέλος μιας εποχής οικονομικού φιλελευθερισμού με τις οικονομικές αγορές ε, ως εχμή του δώρατος της ε, παγκοσμιοποίησης καθώς η ολοκλήρωση των αγορών ήταν πολύ πιο μπροστά από την πολιτική ολοκλήρωση, κάτι το οποίο βεβαίως ήταν σύμφωνο και με το τι συνέβαινε στον υπόλοιπο κόσμο και με τις, ε, το γενικότερο κλίμα. Ίσως αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ νωρί να πούμε το τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι το τέλος μιας εποχής, αλλά δεν ξέρουμε τι ανατέλει ακόμα. Αλλά κάτι που θα έπρεπε να έχουμε κατά νου είναι πως οι πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες των δημοσιονομικών συνεπειών συνήθως έρχονται με διαφορά φάσεις. Και αυτό συμβαίνει και τώρα. Έχω την εντύπωση πως η κρίση μεταξύ άλλων αποκάλυψε ουσιαστικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, έχει αποκαλύψει την αποτελεσματικότητα του δημοσιονομικού, της δημοσιονομικής ρύθμισης, την ανεπάρκεια των διαδικασιών συντονισμού, ειδικά στην Ευρωζώνη, έχει καταδείξει και να στο μηχανισμό επιτήρησης και φαίνεται πως υπάρχει και μία δυναμία από την έλλειψη δυνατότητας ε, δανειστού τελευταίας καταφυγής. Ξέρω πως αυτό το θέμα είναι ακόμα ακαθόδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όσοι βεβαίως συνειδητοποιούν πως νομισματική ένωση χωρίς δανειστή τελευταίας καταφυγής ε, αυξάνονται συνεχώς ο αριθμό αυτών των ανθρώπων. Ποιοι κίνδυνοι τώρα υπάρχουν μπροστά μας. Βεβαίως το δημόσιο χρέος αυξάνεται σε όλα τα κράτη-μέλη και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος του να μην είναι βιώσιμο πλέον αυτό το χρέος. Η δε μεγάλη προσοχή που έχει δοθεί στις διεθνείς αγορές και τα ΜΜΕ στο ελληνικό χρέος ε, έχει μεγάλη σχέση με τη φύση και το μέγεθος της πραγματικής κρίσης στην Ελλάδα αλλά η προσοχή αυτή μας δείχνει και κάτι άλλο πως και τα διεθνή ΜΜΕ και οι διεθνείς χρηματαγορές θεωρούν πως η ελληνική κρίση είναι πρόδρομος άλλων πραγμάτων και το πώς αντιμετωπίζεται η ελληνική κρίση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ενδεικτικό για τον υπόλοιπο κόσμο. Ένας τρόπος βέβαιος είναι η δημοσιονομική σταθερότητα που δεν είναι μόνο επιθυμητό αλλά και απαραίτητο σε πολλές χώρες και ειδικά την Ελλάδα. Αλλά υπάρχει μια λεπτή γραμμή που διαχωρίζει την ε, δημοσιονομική σταθερότητα και την δημιουργία ενός φαύλου κύκλου μέτρων μείωσης ε, του ελλείμματος και αρνητικής ανάπτυξης που θα οδηγήσουν σε βαθία και παρατεταμένη ύφεση που θα μπορούσε να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες όχι μόνο για τις εν λόγω χώρες ε, οικονομικούς και κοινωνικούς όρους αλλά και οικονομικό αντίκτυπο για την υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία. Και πάντα βεβαίως ελοχεύει ο κίνδυνος της απόκλησης των εθνικών οικονομικών τάσεων στην Ευρωζώνη και το ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ε, μη βιώσιμε εξωτερικές ανισορροπίες. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι πως ετέθη ένα ερώτημα τις τελευταίες εβδομάδες που κανείς δεν τολμούσε να θέσει πριν από λίγες εβδομάδες. Δηλαδή το εάν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης στην Ευρωζώνη. Ένα ερώτημα το οποίο λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες πριν δεν τολμούσαμε να θέσουμε. Και κάποιοι ήδη κάνουν συγκρίσεις με την εμπειρία του 92-93 που οδήγησε στην διάλυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Τι πρέπει να γίνει τώρα. Το κατασκεύασμα του Μάστριχ το οποίο προσωπικά συχνά περιγράφω ως ένα μεταμοντέρνο κατασκεύασμα που αψηφά τους νόμους της βαρύτητας και φοβάμαι πως οι νόμοι της ε, βαρύτητας τώρα θα μας εκδικηθούν είναι ένα κατασκεύασμα το οποίο βασίζεται σε έναν πυλώνα μόνο, το νομισματικό, με έναν ασθενή οικονομικό πυλώνα και έναν ανύπαρκτο πολιτικό πυλώνα. Συγκεκριμένα λοιπόν θεωρώ πως πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε στενότερη και δεσμευτική συνεργασία των εθνικών οικονομικών πολιτικών με κίνητρα και κυρώσει ενσωματωμένα, αλλά βεβαίω ε, μπορεί να πει κανείς πως ο συντονισμό ε, είναι εύκολος στα λόγια. Και υπάρχει ένα κρίσιμο πρόβλημα το οποίο θα μας συνοδεύει τους ερχόμενους μήνες, γιατί υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Πώς κατανέμεται το βάρος Τη προσαρμογή μεταξύ των ελληματικών και των πλασματικών χωρών στην Νομισματική Ένωση. Κάποιοι παριστάνουν πως ε, αυτό είναι μόνο ευθύνη των ελληματικών χωρών. Αυτό είναι πολιτικά επικίνδυνο και είναι και λανθασμένα οικονομικά. Χρειαζόμαστε, το δεύτερο που χρειαζόμαστε είναι πιο κοινού και πιο αποτελεσματικού κανόνε συντονισμού για συμπεριλαμβανομένων μέτρων για να ελέγξουμε αυτό το οποίο θα έλεγα πρακτικές καζίνου στις ε, αγορές και μετά χρειαζόμαστε και μηχανισμούς επιτήρησης κατά το οποίο σημαίνει ενίσχυση των εξουσιών της Κομισιόν. Επίσης χρειάζεται ένας δανειστής τελευταίας καταφυγής που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Είναι χρήσιμο, απαραίτητο, αλλά δεν θα γίνει αύριο, γιατί ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε, αλλά κάτι το οποίο είναι απίθανο να συσταθεί του επόμενους μήνες ή και χρόνια, γιατί υποψιάζομαι, μεταξύ άλλων, πως ε, αυτό απαιτεί αναθεώρηση της συνθήκης, κάτι το οποίο δεν θα γίνει αύριο ή μεθαύριο. Οπότε τι χρειαζόμαστε εντωμεταξύ λύσεις ad hoc για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα προβλήματα χωρών όπως η Ελλάδα και πιθανό και άλλων χωρών. Και να προσθέσω δύο πράγματα ακόμα. Πιστεύω πως η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης χρειάζεται μια ενιαία εκπροσώπηση σε διεθνή θεσμικά όργανα και φόρα και θα είναι χρήσιμο και ένα μήνυμα που στον υπόλοιπο κόσμο να ξεκινήσουμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και νομίζω πως χρειαζόμαστε και μεγαλύτερη ανάμιξη των αρχηγών κυβερνήσεων στα της Ευρωζώνης και περισσότερες συνόδους κορυφής της Ευρωζώνης. Βεβαίως όλα αυτά είναι πολλά. Και το ερώτημα του ενός 3 ευρώ είναι το εάν είμαστε έτοιμοι πολιτικά. Εάν είμαστε πολιτικά έτοιμοι για την επόμενη φάση της ΟΝΕ, θα πρέπει να αποτελέσει τίμα μιας ευρύτερης διαπραγμάτευσης για ένα νέο, μια νέα συμφωνία πακέτο που θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα ενίσχυσης εσωτερικής αγοράς, μέτρα μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα και μεταξύ άλλων και αυτό είναι σημαντικό μια ελάχιστη συμφωνία στον συντονισμό εθνικών φορολογικών πολιτικών. Όλα αυτά είναι σημαντικά και φοβάμαι πως δεν έχω χρόνο για το θάρρος να δούμε το επόμενο ερώτημα που είναι το τι γίνεται αν δεν είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη φάση Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα συνεχίσω την... εκεί που σταμάτησε ο Λουκάς Τσουκάλης και θα μιλήσω για τα ίδια μακροοικονομικά θέματα. Θα ήθελα να μιλήσω για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία και θα ήθελα να ξεκινήσω με δύο παρατηρήσεις για το τι έχουμε μάθει ε, κατά την αποψή μου από την κρίση. Ε, το πρώτο σημαντικό μάθημα είναι ότι ένα σύστημα πρόληψης της κρίσης δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε ε, διατάξεις πρόληψης της ε, κρίσης. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε καλούς πυροσβεστήρες και άρα δεν χρειαζόμαστε πυροσβεστική υπηρεσία. Χρειαζόμαστε πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην πρόληψη της κρίσης. Και βέβαια, ε, ένα καθεστώς Πρόληψη τη κρίση δημιουργεί περισσότερου κινδύνους και καθιστά πιο δύσκολη την πρόληψη. Είναι θέμα σχεδιασμού του συστήματος αυτού. Δεν είναι θέμα αρχής. Η, η απλή διάσωση δημιουργεί περισσότερους κινδύνους. Αλλά ένα σύστημα που δημιουργεί περισσότερους, περισσότερες δεν δημιουργεί περισσότερους κινδύνους. Ε, Παραδείγματο χάρη, πηγαίνετε στην Ασία και ρωτήστε τις αν τα, μέσα που τους προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τους δίνουν κίνητρα για να ξαναρχίσουν. Υπάρχει αυτό το θέμα του ηθικού κινδύνου. Ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στην Ευρωζώνη η απουσία ενός συστήματος ε, πρόληψης της κρίσης είναι ε, έλλειψη. Το δεύτερο δίδαγμα είναι ότι κάθε πρόβλημα δεν έχει δημοσιονομική αιτία. Μπορούμε να σκεφτούμε δύο περιπτώσεις που είναι μπροστά μας, η Ελλάδα και η Ισπανία, που έχουμε την Ελλάδα που είναι το πρόβλημά της πιο δημοσιονομικό και την Ισπανία που το πρόβλημά της είναι πιο οικονομικό. Αν δούμε όμως τις υπόλοιπες χώρες, αν δούμε την κατάσταση σε χώρες που έχουν πρόβλημα στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη, ε, και ποιε χώρες δεν έχουν πρόβλημα, θα πρέπει τελικά να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ασθενή σχέση μεταξύ της δημοσομικής διάσταση και της οικονομικής διάσταση. Η προϋπόθεση με την οποία εργαστήκαμε τα τελευταία δέκα χρόνια και όχι μόνο και περισσότερο είναι ότι αν ασχοληθήσεις αν παρακολουθήσεις τον προϋπολογισμό, τα δημοσιονομικά θέματα, επιλύσει τα προβλήματα. Τι υπάρχει από πίσω. Ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι εν γενός ε, σταθερός και ότι οι αιτίε αστάθειας προέρχονται από το δημόσιο τομέα. Αυτό είναι λάθος. Ε, αυτό το μάθαμε από την κρίση και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν δύο ειδών προβλήματα. Τα δημοσιονομικά θέματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, ε, συχνά είναι πηγή αστάθειας, αλλά το γεγονός ότι ελέγχουμε την πηγή αστάθειας δεν σημαίνει ότι ελέγχουμε και όλες τις πηγές αστάθειας. Επομένως, η δημοσιονομική πειθαρχία ή, ή μάλλον η έλλειψη δημοσιονομικής πειθαρχίας δεν είναι η μητέρα όλων των κρίσεων. Επομένως, τι μαθήματα θα πρέπει να μάθουμε πια. Τι θα πρέπει να διδαχθούμε, ούτως ώστε να δράσουμε σωστά για την δημοσιονομική εποπτεία. Θέλω να πω ότι το θέμα που έχουμε μπροστά μας είναι ένα θέμα εφαρμογής κυρίως. Έχουμε ένα σύστημα που υπάρχει, έχουμε το το πιο περίπλοκο σύστημα ε, δημοσιονομικής εποπτείας στην Ευρωζώνη. Έχουμε την νομική βάση, έχουμε τις διαδικασίες, έχουμε τη συνένεση μεταξύ των πολιτικών. Τι λείπει είναι η εφαρμογή. Η περίπτωση της Ελλάδας είναι εμβληματική περίπτωση. Δεν θα την αναλύσω ξανά. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η Κομισιόν όταν παρατήρησε την πρώτη κακή λογιστική της Ελλάδας πρότεινε να ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση. Αλλά α, καθυστέρησε αυτή και κόλλησε στο Συμβούλιο. Ε, δηλαδή υπήρξε μια απόφαση να μην δράσουν. Υπήρχε πρόβλημα εφαρμογής. Δεν είναι πρόβλημα κανόνων. Ήταν πρόβλημα λοιπόν εφαρμογής των κανόνων που ήδη έχουμε. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι ε, μεγαλύτερες ελεκτικές ε, εξουσίες για την Κομισιόν όπως προτάθηκε στις 15 Φεβρουαρίου και αν θέλουμε να σκεφτούμε τι μπορεί να πάει στραβά, ίσως χρειαζόμαστε μια ευρύτερη προσέγγιση πέρα από τα, τις κλασικές για τη δημοσιονομική υποπτία. Ε, γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίες κινούνται πολύ γρήγορα και περνάνε από το δημοσιονομικό πλεόνασμα στο έλλειμμα. Δηλαδή η δημοσιονομική εποπτεία ίσως είναι υπερβολικά απλουστευτική. Έχουμε επικρίνει ε, τις τράπεζες ότι δεν είχαν επαρκή μοντέλα για την αξιολόγηση του κινδύνου. Αλλά αυτά τα, αυτά τα μέτρα, αυτά τα μοντέλα είναι καλύτερα από αυτά που έχουν οι κυβερνήσεις. Δεν έχουμε καθόλου μοντέλα αξιολόγηση του κινδύνου. Και τα μοντέλα είναι δετερμιστικά σε ό,τι αφορά τον καθορισμό του κινδύνου για τους προπολογισμού. Και αν έχουμε σοβαρές καταστάσεις δεν προβλέπουμε τους τι μπορεί να προκύψει. Φυσικά θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τους δημοσιονομικούς θεσμούς και ελπίζω ότι η Ευρώπη να έχει και ελεγκτικές διαδικασίες και εποπτική διαδικασία, ε, διαφορετικές διαδικασίες. Τώρα, η τελική λύση να διώξουμε μια χώρα η οποία δεν συμπεριφέρεται σωστά. Μπορούμε να το σκεφτούμε. Ένα από τα μαθήματα και τα διδάγματα της κρίσης είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε όλα, όλες τις λύσεις. Αλλά η αποτελεσματικότητα σημαίνει κατάλληλες απαντήσεις. Το ΕΚΟΦΗΝ και η Ευρωζώνη δεν είχαν τη θέληση να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία. Ε, για τη διαχείριση της κρίσης. Το δεύτερο, ο δεύτερος άξονας που θέλω να αναλύσω εδώ. Όπως είπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργό, η Ελλάδα έχει ένα πρόγραμμα τύπου Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Και αν ήταν εκτό της Ευρωζώνης θα είχε στραφεί προς το διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως η Ουγγαρία και άλλες χώρες. Η Ελλάδα δεν είναι επιλέξιμη για βοήθεια εξαιτία του άρθρου 143 που λέει ότι η βοήθεια δίδεται σε χώρες με μια παρέκκληση. Υπάρχει λοιπόν ε, δυνατότητα βοήθειας εκτός της Ευρωζώνης, όχι εντός της Ευρωζώνης όμως. Το θέμα είναι γιατί. Υπάρχει μια σύγχυση πνευματική νομίζω μεταξύ δύο πραγμάτων. Απ' τη μία είναι η αρχή της μη συνυπευθυνότητας ε, του δημόσιου χρέους. Άρθρος 125. Αυτό είναι θεμελιώδης αρχή του ευρώ και θα πρέπει να παραμείνει. Είναι ένας βασικός πυλώνας. Δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητήσουμε καθόλου αυτή την αρχή. Η άλλη αρχή είναι ότι δεν υπάρχει βοήθεια. Η αρχή της μη βοήθειας. Δεν δίνουμε δάνεια δηλαδή για να βοηθήσουμε μια χώρα που ανήκει στην Ευρωζώνη. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Όταν το Διεθνές δομισματικό Ταμείο δίνει βοήθεια δεν παίρνει την ευθύνη για το χρέος αυτής της χώρας. Δίνει βοήθεια και δάνεια και κερδίζει και λεφτά από αυτό. Επομένως αυτές οι δύο αρχές δεν είναι καθόλου ταυτόσιμες. Αλλά κάπως, κάπως έγινε και σκεφτήκαμε ότι είναι ταυτόσιμες. Εγώ νομίζω ότι είναι εντελώς εσφαλμένο αυτό. Είναι μια διανοητική σύγχυση, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε και να εφαρμόσουμε το άρθρο 125 και ταυτόχρονα να υπάρχει βοήθεια υπό όρους. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι λοιπόν ε, για αυτά τα θέματα πριν οποιαδήποτε συζήτηση. Αν πιστέψουμε, αν ε, θεωρήσουμε ότι υπάρχει χώρος για βοήθεια, υπάρχουν δύο συν μία, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, ε, το κλασικό καθεστώς ε, των δανείων και τρίτη λύση, ο συνδυασμός των δύο που υπάρχει σε πολλές μη ευρωπαϊκές χώρες. Με ένα συμπεφωνημένο πλαίσιο που θα είναι ιδιάζων για την Ευρωζώνη. Αυτή λοιπόν είναι η λύση. Θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε μια σαφή επιλογή και πρέπει να έχουμε ένα σύστημα βοήθειας υπό όρους που να μπορεί να λειτουργήσει στο μέλλον. Τέλος, υπάρχει ένα τελευταίο θέμα, η μεταρρύθμιση του καθεστώτος οικονομικής εποπτείας. Το θέμα δηλαδή της ανταγωνιστικότητας του ισοζυγίου τρεχουσών πληρωμών. Αυτό είναι ένα μη δημοσιονομικό θέμα. Θα πρέπει να το δούμε χωριστά. Έχουμε νομική βάση, το άρθρο 121. Υπάρχει το νέο άρθρο 126. Δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν νομικής βάσης. Υπάρχει πρόβλημα ότι δεν υπάρχει μία συμφωνία για αυτή την εποπτεία. Ένας ομιλητής είπε προηγουμένως, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε το ισοζύγιο τρεχουσών πληρωμών. Δεν συμφωνώ. Οι, τα ισοζύγια τρεχουσών πληρωμών δείχνουν πού μπορεί να κοίτονται οι κρίσεις. Αλλά δεν είναι από μόνο τους προβλήματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα ελλείμματα ή τα πλεονάσματα ε, του ισοζυγίου τρεχουσών πληρωμών πάνω από ένα εκατό είναι, είναι το πρόβλημα. Μπορούμε να πούμε βεβαίως ότι όταν εξεπράνει το 10% του ΑΕΠ είναι πρόβλημα. Αλλά βεβαίως αυτό από μόνο του δεν δίνει απάντηση στο ερώτημα. Το θέμα είναι τι υπάρχει από πίσω. Υπάρχουν επενδύσεις, υπάρχει κατανάλωση, είναι ανάπτυξη λόγω των ακινήτων. Δεν υπάρχει λοιπόν καθολική, καθολικό benchmark μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, ως δείκτη το ισοζύγιο τρεχουσών πληρωμών και να αξιολογήσουμε την κατάσταση ε, και με όρου ανταγωνιστικότητα. Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα έχουμε οπισθοχωρήσει. Γιατί τη στιγμή του ERM υπήρχε μια σοβαρή συζήτηση για τι αναλυματικέ ισοτιμίε, για την ανταγωνιστικότητα. Τώρα φτάσαμε σε μια κατάσταση όπου δεν μιλάμε ε, για την ονομαστική αλλά για την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία τα ίδια ουσιαστικά προβλήματα υπάρχουν. Υπάρχουν πολιτικές που μπορεί να αυξήσουν τους φόρους και μπορεί να μειώσουν την κοινωνική προστασία. Αυτό θεωρείται υποτίμηση, αλλά θεωρείται φορολογική πολιτική. Δεν το συζητάμε γιατί είναι κυρίαρχο τομέα των κρατών μελών. Αλλά στην πράξη είναι υποτίμηση. Επομένω, όλα θα πρέπει να συζητηθούν, όλα θα πρέπει να τεθούν επιτάπητο. Χρειαζόμαστε λοιπόν διαδικασίε για να ξεκινήσουμε σοβαρέ συζητήσει. Μία συστηματική δηλαδή ε, εποπτεία των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Και να βάλουμε εδώ και μία πολυμερή διάσταση. Ε, συζητάμε το θέμα της συμμετρίας ή ασυμμετρίας ε, να χρησιμοποιήσουμε τα νέα εργαλεία. Το άρθρο που λέει ότι υπάρχουν πολιτικές που μπορεί να θέσουν ένα αμφιβόλο την ε, νομισματική ένωση και αυτές θα πρέπει να εμποδιστούν. Θα πρέπει να υπάρξει τροχοπέδι σε αυτές τις πολιτικές. Υπάρχει χώρος δράσης λοιπόν. Υπάρχει δυνατότητα η Ευρωζώνη επίσης να δράσει. Δημιουργήθηκε ως ο θεσμός που αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτά τα προβλήματα, αλλά δεν έκανε τίποτα στην κρίση. Ήταν απογοήτευση. Το θέμα είναι πώς θα δικοδομήσουμε συνένεση, πώς θα δράσουμε. Το έγγραφο το οποίο δημοσιεύτηκε την Δευτέρα από την Ευρωζώνη είναι ε, ευπρόσδεκτο. Και επιπλέον οι κυβερνήσεις βεβαίως θα πρέπει να προχωρήσουν με τα κατάλληλα εργαλεία. Η ανταγωνιστικότητα είναι με, μείζον μέλημα. Δεν μπορούμε να μην έχουμε τα εργαλεία να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Βέλγιο παρακολουθεί τις ε, ε, εξελίξεις των μισθών και προσπαθεί το Βέλγιο η ανάπτυξη και η εξέλιξη των μισθών να μην υποσκάψουν την ανταγωνιστικότητα. Όλη αυτή η συζήτηση που μας περιμένει νομίζω ότι είναι και συζήτηση όπου το Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει ένα σημαντικότατο ρόλο. Thank you very much, Chairman. It's an honor to be here. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είναι τιμή μου που είμαι εδώ και δεν θέλω να μιλήσω τελευταία, δεν είναι εύκολο μετά από αυτές τις παρουσιάσεις. Αυτό το οποίο θα κάνω εγώ στα 17 λεπτά είναι να εξετάσω ειδικά τις ε, κρατικές δομές και θεσμικά όργανα καθώς και τα κίνητρα που υπάρχουν ε, αυτή τη στιγμή σε συνδυασμό με την ε, οικονομική διακυβέρνηση όπως την έχουμε δει τελευταία χρόνια αλλά και το ποιες μεταρρυθμίσεις μπορούν να γίνουν. Να ξεκινήσω με μια σύντομη περιγραφή των ελλείψεων της διακυβέρνησης της ΟΝΕ. Της έχω βάλει σε τρεις κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα διαχείριση κρίσεων, επιτήρηση και συντονισμός και τρίτον ζητήματα νομοποίησης. Όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, νομίζω πως η Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο και άλλα βήματα το έχουν αναλύσει αυτό το θέμα σε 10 χρόνια που έχουν περάσει από την ΟΝΕΟ, οπότε θα είμαι σύντομη. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα πως ο συντονισμός δημοσιονομικών κυρινήτρων δεν επαρκεί και αυτό το οποίο έχουμε δει είναι τα, ενδιαφέροντα, τα εξή ενδιαφέροντα στοιχεία. Δεν έχουμε σκεφτεί μία δημοσιονομική στάση που θα είναι κοινή σε ολόκληρη την ΟΝΕ δεν υπήρχε ρόλο τη ε, Κομισιόν και δεν υπάρχει και αρκετά μεγάλη ευελιξία του κοινοτικού προπολογισμού. Και βεβαίω η εμπειρία του παρελθόντος ε, θέτει ερωτήματα και για το τι θα γίνει στο μέλλον και για μια στρατηγική εξόδου. Δεύτερο μεγάλο στοιχείο είναι βεβαίω η κρίση του δημοσίου χρέους. Το έχουμε συζητήσει στι προηγούμενε παρουσιάσει και θα συμφωνούσα με τον προλαλήσαντα συνάδελφο έχουμε δει πως υπάρχουν ε, κάποιες ε, δομές ε, οι οποίες είναι λανθασμένες όσον αφορά τα κίνητρα και τα εργαλεία δεν επαρκούν για να διαχειριστούμε τη ρευστότητα και το πρόβλημα της φερεγγιότητας. Δεν υπάρχει επίσης αρκετή πειθαρχία. Επίσης η πιθανότητα του να αφήσουμε μια χώρα να προχωρήσει σε στάση πληρωμών ή να βγει από την ΟΝΕ δεν υπάρχουν ως τελευταία λύση. Δεν Υπάρχει επίσης μία κανονική διαδικασία στάση πληρωμών ενός κράτους, ούτε ένας δανειστής τελευταίας καταφυγής. Τώρα, εγώ δεν θα μιλήσω για την επιτήρηση των χρηματαγορών. Θα αναφερθώ στην επιτήρηση και συντονισμό δημοσιονομικής πολιτικής και οικονομικής πολιτικής. Πρώτα απ' όλα νομίζω πως υπάρχει μία έλλειψη αξιοπιστίας ε, του Συμφώνου Σταθερότητας ε, και Ανάπτυξης γιατί σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη παρουσιάζουν το, παραβιάζουν το 3% αλλά και γιατί υπάρχει έλλειψη δεσμεύσεων να επιστρέψουμε στα απαιτούμενα επίπεδα και, και οι δεσμεύσει αυτέ που έχουν αναλυφθεί δεν είναι πάρα πολύ αξιόπιστε. Επίση, όσον αφορά την οικονομική πολιτική και συντονισμό, δεν έχει αναλυφθεί δράση όσον αφορά τι αποκλήσει στην ανταγωνιστικότητα και στο ισοζύγιο τροξών συναλλαγών. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι γνωστά τα δεδομένα εδώ και χρόνια και αυτό είναι αποτέλεσμα και της κρίσης λόγω πολλών προβληματικών χωρών αλλά το γεγονός πως έχουμε αυτές τις αποκλήσεις οδήγησε στην εξή κατάσταση. Ο αντίκτυπος της κρίσης είναι χειρότερος από ό,τι θα ήταν αλλιώς. Και βλέπουμε πως τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα δεν έχουν επιληθεί και στις χώρες και στην εσωτερική πολιτική συζήτηση βλέπουμε πως δεν ξέρει πως να το αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και Τρίτον, για τον συντονισμό είναι το πρόβλημα του κατά πόσο είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο, καθώς κάποιοι θεωρούν ότι είναι εσωτερική υπόθεση. Δεν ξεκίνησε τώρα με τις προτάσεις αυτές, ξεκίνησε πριν από 9 χρόνια, όταν η πρώτη χώρα κατονομάστηκε η Ιρλανδία δηλαδή υπό τις ε, τότε κατευθυντήριες γραμμές και υπήρχε η αίσθηση πως ο μηχανισμός δεν λειτουργεί και πως το να κατονομάσουμε μια χώρα δεν σημαίνει και πως ε, συνεργάζεται και έκτοτε βεβαίως ε, η διαδικασία συντονισμού αυτή παραμένει στα χαρτιά και βεβαίω είναι και το ζήτημα του πώς θα γίνει αποδεκτό ένα τέτοιο πολιτικό αποτέλεσμα στο συνολικό επίπεδο της ΟΝΕ και το εάν ε, μεμονωμένες χώρες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα εκτός της ΟΝΕ οπότε είναι ζητήματα που θα πρέπει να τα ξαναδούμε στο μέλλον οι αιτίε για όλες αυτές τις ελλείψεις τώρα θα τις ε, περιέγραφα ως εξής. Έχουμε ένα ατελές ε, πλαίσιο θεσμικό και λειτουργικό το οποίο έχει λίγο μεταρρυθμιστεί από την συνθήκη του Μάστριχτ. Αν και έχουν γίνει κάποια βήματα, π.χ. και το σύμβουλο Σταθερότητα και Ανάπτυξη μετά το Μάστριχτ και μετά μεταρρυθμίστηκε, δημιουργήθηκε το Eurogroup και αυτό έχει μεταρρυθμιστεί. Τώρα υπάρχει πρόεδρος, αναφέρεται συνθήκη κτλ και είχαμε και την πρώτη σύνοδο κορυφή Ευρωζώνης, αλλά εγώ δεν θεωρώ πώ θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ πέρα. Έχουμε την εμπειρία 11 ετών ΟΝΕ και την κρίση. Δεύτερον, δεν έχουμε αντιληφθεί την πραγματικότητα της ε, ΟΝΕ, ότι όλοι μαζί είμαστε στην ίδια βάρκα. Οι περισσότεροι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι στα εθνικά ΜΜΕ, αν διαβάσουμε τα σχόλια π.χ. για την ε, συνθήκη της, ε, που υπογράφουν οι δύο κυβερνητικοί εταίροι. Έχουν την αίσθηση πως καθορίζουν τελείως ε, την οικονομική τους πολιτική. Δεν έχουν αντιληφθεί ούτε το κοινό ούτε η πολιτική. Το ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τη μακροοικονομική ανάλυση. Δεν το έχουν λοιπόν αντιληφθεί αυτό. Και τέλος ε, όσον αφορά το πώς ελέγχονται και βεβαίως το ότι είναι εθνικές οι εκλογές βεβαίως δεν έχουν κανένα κίνητρο οι πολιτικοί να συμπεριφέρονται σωστά ως προς την ΟΝΕ. Ναι». Αλλά υπάρχει λοιπόν ένας κίνδυνος, ε, προβλήματα μονοθετικού κινδύνου και υπάρχει και το συνεχές ε, πρόβλημα ότι δεν υπάρχει συνεργασία αν και θα μπορούσε να είναι αμοιβαία αποφελής. Τέλος ο ρόλος ε, υπερεθνικών φορέων, ειδικά της ε, Κομισιόν, στην προώθηση της ε, ΟΝΕ ναι, έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Και αυτό οφείλεται και στα κράτη-μέλη, τα οποία στο παρελθόν προσπάθησαν να περιορίσουν την υπερεθνική διάσταση σε πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό π.χ. παραδείγματο χάρη αφορά τον συντονισμό του κινήτρου ή π.χ. τις εξής Eurostat που εδώ και 6-7 χρόνια σέρνονται και βεβαίω το πώς θα κατανομάζουμε και θα το πιάσουμε διάφορα και Συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο να υπάρξει μια ευρωπαϊκή λογική γιατί υπάρχει ένα σημαντικό ρόλο στην νομοθετική διαδικασία αυτή τη στιγμή που μόλις τώρα τον ανακάλυψαν οι εθνικές κυβερνήσεις και υπάρχει και η πολιτική ουσία που μπορεί να διατυπωθεί από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ζητήματα που δεν είναι στη συναπόφαση τώρα να αναφερθώ στο πολιτικό πλαίσιο της διακυβέρνησης ΟΝΕ σε τρία επίπεδα. Πρώτα απ' όλα το πλαίσιο της ΟΝΕ, το πλαίσιο των εθνικών κυβερνήσεων και την κατάσταση στο εσωτερικό. Θεωρώ πως εδώ πέρα υπάρχει ένα παράθυρο, μια στιγμή ευκαιρίας Πρώτα απ' όλα υπάρχει η οικονομική και η κοινωνική και δημοσιονομική κρίση, περίπτωση της Ελλάδας και δύο συζητήσεις ε, που σχετίζονται. Πρώτα απ' όλα η στρατηγική 2020 και η συζήτηση για τον προπολογισμό. Βλέπουμε όμως πως υπάρχει εστίαση στην διαχείριση και πρόληψη του κινδύνου και μικρές φιλοδοξίες για να υπάρξει περισσότερη κοινή οικονομική πολιτική. Η έμφαση λοιπόν μάλλον είναι στην Ελλάδα και όχι στη στρατηγική του 2020. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αντιμετωπίσει ζητήματα οικονομικά και δημοσιονομικά. Υπάρχει η σύνοδο στις 11 Φεβρουαρίου, θα υπάρξει άλλη μία το Μάρτιο και θα είναι και στην σύνοδο του Ιουνίου. Αλλά τι γίνεται με την προοπτική της ΟΝΕ. Κατά την άποψή μου υπάρχει ένας κίνδυνος ότι λόγω της ε, ιδέας, ότι λόγω της ιδέας του ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια οικονομική κυβέρνηση, που βεβαίως δεν είναι άξια του ονόματος, δεν ε, χρειάζεται κάποιο παραπάνω μέτρο για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της ΩΝΕ. Τώρα, τι ε, χρειάζεται στο πολιτικό πλαίσιο. Βέβαια, εγώ εργάζομαι στο γερμανικό πλαίσιο, οπότε ίσως έχω επηρεαστεί από αυτό. Υπάρχει λοιπόν απροθυμία να αποδεχτούν περισσότερη παρέμβαση από το ευρωπαϊκό επίπεδο πλην κρίσεων. Αυτό φαίνεται και από τις θέσεις για τη στρατηγική για την ε, Ένωση 2020, π.χ. όταν μιλάμε για συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, μηχανισμούς συντονισμού και τις ε, θέσεις βεβαίως ε, για το τι θα γίνει με την ε, θέση των κυβερνήσεων στην νομοθετική διαδικασία. Οπότε, μακροπρόθεσμα δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση συντονισμού. Πλην τη Ελλάδα, βέβαια, γιατί όλοι εδώ πέρα συμφωνούν. Επίσης, θα έλεγα πως υπάρχει ένα πλαίσιο όπου υπάρχει ο κίνδυνος ε, στι χώρε εκείνες που θεωρούν ότι πληρώνουν ε, συνεχώς μπορούμε να δούμε ότι θα μεταβληθεί η άποψη για τον βαθμό αλληλεγγύης και συνοχής που απαιτείται στην ΟΝΕ. Και βέβαιως θα υποχωρήσουν αυτές οι αντιλήψεις, κάτι το οποίο είναι προβληματικό. Τώρα όσον αφορά το εσωτερικό πλαίσιο, θεωρώ πως η ανταγωνιστική πίεση και η ανάγκη πραγματικής υποτίμησης που αφορά πολλά κράτη μέλη μπορεί να έχει πολιτικό αντίθετο τα επόμενα χρόνια για πολλές χώρες υπάρχει ο κίνδυνος πολιτικού κατακερματισμού, λαϊκισμού στα άκρα, κάτι το οποίο μπορεί να εξασθενήσει την όρεξη κυβέρνησης για μακροπρόθεσμα έργα ολοκλήρωσης, οπότε εδώ πέρα υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος και βεβαίω υπάρχουν και συνταγματικά εμπόδια στην περαιτέρω ολοκλήρωση, όπω π.χ. στη Γερμανία. Αυτό είναι ουσιαστικό, αλλά είναι και ένα πολιτικό επιχείρημα, βέβαια, για να αποφευθεί περαιτέρω συζήτηση. Τέλο θα έπρεπε να ανησυχούμε για τι εξελίξει κοινή γνώμη. Αν δούμε την ιστορία τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. υπάρχει σαφή σχέση μεταξύ τη υψηλή ανεργία, χαμηλή ανάπτυξη και τη χαμηλή υποστήριξη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό το είδαμε και στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80. Και αν αναμένουμε τέτοιες εξελίξεις το 2010 και 2011 κοινωνικές εντάσεις και τα λοιπά, θα πέσει η στήριξη προς την ενοποίηση. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως από την άλλη είναι πως οι πολίτες έχουν περισσότερες προσδοκίες όσον αφορά τη δυνατότητα της Ένωσης να λύσει προβλήματα σε κοινωνικά και οικονομικά επίπεδα. Κάτι το οποίο βεβαίω είναι θετικό, αλλά περιέχει και τον κίνδυνο τη απογοήτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και του εθνικού πολιτικού. Οπότε το συμπέρασμα είναι πω έχει περισσότερη σημασία η επικοινωνία και η ηγεσία για τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ και για τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Ε, ο χρόνος μου τελειώνει. Οπότε θα ήθελα να τελειώσω με δύο διαφάνειες ε, για τις προτεραιότητες για την ΟΝΕ, διακυβέρνηση, μεταρρύθμιση. Πρέπει να επιταχυνθεί η παρακολούθηση, πρέπει να μεταρρυθμιστεί το σύμφωνο σταθερότητας. Εγώ θα αξιολογούσα την δήλωση του Eurogroup της περασμένης εβδομάδας, όπου για πρώτη φορά ε, αναφέρθηκε η ανάγκη ανισορροπιών και το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, είναι κάτι σημαντικό εφόσον συμφώνησε και η γερμανική κυβέρνηση, αλλά το πώς θα πιεστούν οι κυβερνήσεις για να ακολουθήσουν το άρθρο της συνθήκης για ζητήματα που λέει ότι είναι κοινά, είναι κάτι ανοιχτό. Εγώ θα έλεγα πως θα πρέπει να μπλακούν τα εθνικά κοινοβούλια εδώ πέρα σε ζητήματα, ναι. Τώρα, η Ελλάδα πολλά υπόθηκαν για την Ελλάδα, δεν θα πω τίποτα άλλο. Όσον αφορά τις θεσμικές εξελίξεις ε, της ΟΝΕ, ναι, πρέπει να έχουμε κατά νου πως πρέπει να έχει δικε της, δικές της θεσμικές δομές και κάποιον συντονισμό. Εγώ θα έλεγα πως χρειάζονται περισσότερες ε, σύνοδοι κορυφής Ευρωζώνης μαζί με την Ιαρινή Σύνοδο το εάν ε, χρειάζεται το Eurogroup και σε άλλους σχηματισμούς Συμβουλίου. Η στρατηγική του 2020 και ο προπολογισμό ε, πρέπει να έχουν μια συνεκτική αντιμετώπιση, κάτι το οποίο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή και θα τελειώσω, τελειώνω. Πρέπει να δούμε και αυτή την πολιτική απόκληση για να ενισχυθεί το Eurogroup. Για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία η Γαλλία και η Γερμανία να είναι υπεύθυνε για τις εθνικές στρατηγικές τους και να τονίσουμε τη σημασία αυτών των δύο χωρών που μαζί έχουν το 50% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Λοιπόν, πρέπει να έχουν κοινό βήμα. Ευχαριστώ. Äh, ε, και περνάμε στον επόμενο, στο γύρο των ερωτήσεων. Ξεκινάμε με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό ε, Κόμμα. Ποιο ε, από τους συντηρητικού θέλει να κάνει ερώτηση. Κανεί Περνάμε λοιπόν στην Περβάνο Σουμπερέ. Α, Ελίζα. Πρώτα η Ελίζα. thank you very Ευχαριστώ για τις ε, παρουσιάσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες γιατί πήγαν σε μεγαλύτερο βάθος. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Αφορά δύο βασικούς τομείς. Ας προσπαθήσουμε να δούμε Ποιε είναι οι περιοχές, ε, οι βέλτιστες περιοχές νομίσματος ε, και πώς μπορούμε να έχουμε μια βιώσιμη νομισματική ένωση. Μια συζήτηση που είχε γίνει ε, στο παρελθόν και οι προποθέσει. Αυτό ξεχάστηκε από τι συζητήσει μας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα επανέρχεται. Επειδή μιλάτε για την διαφορετική διαφοροποίηση των οικονομιών, νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το σημείο. Τώρα, στην πράξη αν έχουμε διαφορετικά επίπεδα ανταγωνιστικότητας, θα είναι πολύ δύσκολο να επιζήσουμε σε έναν ε, παγκοσμιοποιημένο κόσμο ε, και με τις πηγές ανταγωνισμού που έχουμε τώρα. Πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε τώρα, πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τις ε, πολιτικές συνοχής στα νέα δεδομένα. Όλα αυτά βεβαίως εντάσσονται στην προσέγγιση που ανέφερε ο τελευταίος ομιλητής, δηλαδή αν υπάρχει η πολιτική βούληση να κάνουμε κάποια πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να προχωρήσετε λίγο τον προβληματισμό προς αυτή την κατεύθυνση. Τα διαφθορτικά ταμεία ε, που δημιουργήθηκαν το 1970 είναι το βασικό ε, εργαλείο συνοχής σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Μπορούμε να παραμείνουμε σε αυτά μόνο θέλουμε να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικότητα με βάση την καινοτομία και τις ε, δεξιότητές μας. Μπορούμε να παραμείνουμε λοιπόν σε αυτή τη λογική του 70. Να ακούσουμε τρεις ερωτήσεις και μετά να απαντήσουν οι ομιλητές μας. Η κυρία Αλβάρε. Συγγνώμη κυρία Σβάρτσερ αν δεν προφέρω καλά το όνομά σας, αλλά εδώ μας έχετε ρίξει το γάντι όταν είπατε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό όραμα και όχι μία ατομική εθνική άποψη. Όμως ε, στην ε, κρίση τι γίνεται, ζητάνε από τα κράτη-μέλη μεμονωμένα να αναλάβουν τις προσπάθειες και αυτό θα έπρεπε και ρωτώ δηλαδή, ε, ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να καταλήξουμε σε αυτό που είπε ο κύριος Παπανδρέου, δηλαδή πώς θα έχουμε παραπάνω Ευρώπη ούτως ώστε... οι χώρε να μπορέσουν να ξεπεράσουν την κρίση και ποια μέσα έχουμε στη διάθεσή μα για να ολοκληρώσουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ και τους ε, τρεις ε, που μας κάνατε ολοκληρωμένες παρουσιάσεις ε, αλλά και γιατί πραγματικά ήσασταν μετριοπαθείς, σταθμισμένοι σε αυτά που είπατε. Ε, πολλές φορές η Ευρωζώνη στέλνει βία μηνύματα τα οποία δεν είναι πολλές φορές ανάλογα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει μένει οι ΔΕ. Εγώ δεν είμαι ακόμη καθαρή στις ιδέες μου για την οικονομική επιτήρηση. Λέτε εσείς το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει πράγματα. Αλλά πώς το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει κάτι συνδυάζοντας ε, την ε, γερμανική άποψη με την ελληνική άποψη. Τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο ούτως ώστε να προχωρήσει το πακέτο εποπτείας το οποίο εξετάζεται σήμερα στο Κοινοβούλιο Μιλήσατε εσείς για σταθερότητα και δεν χρειάζεται μόνο δημοσιονομική ε, σταθερότητα αλλά γενικότερη σταθερότητα, οικονομική σταθερότητα. Μπορεί να περάσει αυτό το μήνυμα και στη Γερμανία ότι αυτή η σταθερότητα μπορεί να μας οδηγήσει να αποφύγουμε την κρίση αύριο Ποιο είναι λοιπόν το επιχείρημα, γιατί ξέρω ότι θα δοθεί μάχη στο Συμβούλιο. Για την ελληνική κρίση πολλοί λένε μερικά πράγματα, αλλά μετά μπορεί να αναλάβουν ακριβώς την αντίθετη θέση όταν θα μιλήσουν για τα παράγωγα ή για τα ΣΒΑΠ κλπ. Ευχαριστώ. Καταρχάς, όπως ξέρετε, έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια για το αν η Ευρωζώνη μοιάζει σαν μια βέλτιστη περιοχή νομίσματος ή όχι. Και ξέρετε ότι οι διάφορες οικονομίες το έχουν συζητήσει. Η τάση είναι ότι μια τέτοια περιοχή βέλτιστη νομίσματος θα δημιουργηθεί εν συνεχεία. Αλλά δεν θα προϋπάρχει βέβαια. Αυτό προϋποθέτει ότι οι πολιτικές θα υιοθετηθούν με ένα τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε να, οδηγήσουν σε μια ε, αυξανόμενη σύγκληση των ε, διεθνών οικονομικών τάσεων. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο τα τελευταία χρόνια. Ζήσαμε με την αυταπάτη για 10 χρόνια ότι όλα ήταν καλά, γιατί, για να χρησιμοποιήσω και την έκφραση του συναδέλφου μου, ε, ήταν η περίοδος ε, των παχιών αγελάδων. Ε, τώρα τέλειωσε αυτή η περίοδος. Και κάποια από τα θεμελιώδη που χρειαζόμαστε ε, για να ζήσουμε καλά δεν υπάρχει. Ε, έχουμε ε, και ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών πληρωμών, έχουμε ανεξέλεγκτα ελλείμματα του προπολογισμού κτλ. Έχουμε προβλήματα με τη σύγκληση. Μας επικρίνατε. Ή μάλλον είπατε γιατί δεν θέσαμε το θέμα των πολιτικών συνοχής και των ταμείων συνοχής. Δεδομένης της σημερινή κατάστασης και δεδομένης της ευαισθησία που έχει δημιουργηθεί για αυτές τις ε, ad hoc ρυθμίσεις για να αντιμετωπίσουμε την ελληνική κρίση αλλά και άλλες θα ήταν υπερβολικά πολύ να θέσουμε και θέματα αναδιανομής του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι αυτό έχει περισσότερο πολιτική χρειά. Ειλικρινά σας λέω όμως, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα για μια ριζική επανεξέταση του στοιχείου της συνοχής στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Η πολιτική θέληση δεν υπάρχει για να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι κρίμα κατά την άποψη πολλών, αλλά έτσι είναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική, τις δημοσιονομικές ρυθμίσεις και τους δημοσιονομικούς κανόνες. Ξέρετε ότι η χρηματοπιστωτική κρίση ήταν η αρχή της κρίσης. Ήταν το α. Τώρα περάσαμε από επιδρομές ε, στις τράπεζες στα, σε επιδρομές στα κράτη. Και τα επόμενα, τους επόμενους μήνες και χρόνια θα έχουμε περισσότερες τέτοιες επιδρομές σε κράτη. Θεωρούσαμε ότι η χρηματοπιστωτική κρίση δημιούργησε την απαραίτητη πολιτική βούληση για μια νέα ριζοσπαστική προσέγγιση στην, ε, στις χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις. Αλλά τώρα ξαφνικά ο κόσμος μετά από μερικούς μήνες το ξανασκέφτεται και είναι διστακτικό. Υπάρχουν μερικές τάσεις ε, σε ορισμένε χώρες και σε, σε ορισμένε πολιτικές οικογένειες να τα ξεχάσουμε όλα. Να ξαναμπούμε ας πούμε στο χορό σαν να μην τρέχει τίποτα. Θα ήταν τραγικό κάτι τέτοιο. Γιατί θα, ξανα... θα ξαναδούμε σε λίγο την επόμενη κρίση η ελληνική κρίση ε, εστίασε το πρόβλημα στο CDS, τη Συμφωνία ανταλλαγή Κινδύνων. Ε, αυτό το θέμα δεν είναι διαφανές θέμα, δεν είναι μια διαφανής αγορά. Και το λέω γενικά. Ε, δίνει τη δυνατότητα λαθροχειριών, χειραγωγήσεων και υπάρχουν πολλές δυνατότητες να κερδοσκοπήσει πολύ γρήγορα κάποιος σε αυτό το χώρο. Ε, ελπίζω τώρα, νομίζω φαίνεται ότι υπάρχει μια πολιτική βούληση, όλο ένα και πιο μεγάλη για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και ελπίζω να υπάρξουν και συγκεκριμένα μέτρα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Λέει για την, την περιοχή βέλτιστου νομίσματος. Συμφωνώ με την απάντηση του Λουκά και θέλω να προσθέσω δύο πράγματα. Καταρχάς, η ολοκλήρωση των αγορών είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει ε, στην καλύτερη λειτουργία της Ευρωζώνης. Ε, τα κανάλια ανταγωνιστικότητας μέσω των οποίων οι διαφορές στις, ε, στην ανταγωνιστικότητα διορθώνονται μέσω των δυνάμεων της αγοράς δεν είναι επαρκή. Το να ολοκληρώσουμε περισσότερο τις αγορές μπορεί να βοηθήσει για να ενδυναμώσουμε αυτό το κανάλι που είναι εκ των όνου κάνευ για τη λειτουργία της Ευρωζώνης. Αυτό συνδέει την, το θέμα του ενιαίου νομίσματος με τις ενιαίες αγοράς. Γι' αυτό πρέπει να συμπληρωθεί και με πολιτικές και με εποπτεία. Το τόνισε αυτό. Για τις πολιτικές. το ερώτημα που θέσατε. Έχω την αίσθηση και εγώ όπως ο Λουκάς ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν υπάρχει βούληση και όρεξη για μεγάλες πρωτοβουλίε. Επομένως, η ατζέντα τι θα είναι. Να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε με τον καλύτερο τρόπο και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που είναι μπροστά μας. Η ικανότητα να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες συνέπειες της κρίσης καθώς εμφανίζονται είναι ένα, θα είναι ένα βασικό στίχημα για να επιβεβαιωθεί η νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν φτάσουμε τα όρια, έχοντας χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχουμε, τότε μπορεί να ακουστεί το επιχείρημα να πάμε πιο πέρα. Αλλά πρέπει πρώτα να φτάσουμε στο όριο αυτό. Δεν το έχουμε φτάσει ακόμα. Ας φτάσουμε σε αυτό το χαράκομα και τότε θα δούμε αν υπάρχει άλλη δυνατότητα για κάτι άλλο. Τώρα. Πιστεύω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διότι η μακροοικονομική επιτήρηση και η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση και εδώ όταν μιλάμε για την ε, κατάσταση στην Ισπανία μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με το άρθρο 121 και τα μακροοικονομικά μέσα που μας δίνει και μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε επίσης με αυτά τα μακρο... την μακροπροληπτική εποπτεία στο μέλλον. Όμως το θέμα είναι τι κάνουμε συγκεκριμένα. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν με μακροπροληπτικά μέσα που θα μπορούσε κανείς ε, να λύσει το θέμα ε, της κρίσης όπως προέκυψε από την ε, πολιτική των ακιδίτων. Αν εμείς περιοριστούμε μόνο στην επιτήρηση, στην τραπεζική επιτήρηση, δεν πρόκειται να πάμε μακριά. Πολλές φορές ε, τα τραπεζικά συστήματα εξαρτώνται από εξωτερικές τράπεζες, οπότε το θέμα ενίκο και το τραπεζικό πρόβλημα είναι πράγματα εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, ναι. Ναι, ευχαριστώ. ευχαριστώ μία λέξη μόνο. Συμφωνώ με όλα όσα ακούστηκαν και για μένα η ατζέντα της Ενίας αγοράς προφανώς πρέπει να συνδεθεί με τις σκέψεις αυτές για την ΟΝΕ. Πρώτα απ' όλα το πρόβλημα του κατά πόσο είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο στο εσωτερικό δηλαδή να υπάρχει μια ατζέντα της Ενίας αγοράς που για κάποιες χώρες τουλάχιστον θα πρέπει να συνοδευτεί από, μια, από ένα κοινωνικό πρόγραμμα γιατί νομίζω πως η αποδεκτότητα μεταρρυθμίσεων της εσωτερική αγοράς που θα είναι μόνο απελευθέρωση δεν θα είναι πολύ μεγάλη σε πολλές ε, χώρες. Δεύτερον, εάν προχωρήσουμε παραπέρα μετά της ε, ιδανικής ε, περιοχής ενός νομίσματος υπάρχουν και πολιτικά κριτήρια βεβαίως τουλάχιστον της ε, τελευταίας μορφή. Και ε, μπορούμε να δούμε πως οι δημοσιονομικοί μηχανισμοί θα έλεγαν κάποιοι πως ε, δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες γιατί δεν υπάρχει ένας μηχανισμός δημοσιονομικής θεροποίησης. Εξού και μεγάλη διαφορά μεταξύ Ευρωζώνης και ΕΠΑ όπου λειτουργούν οι αγορές διασυνοριακά καλύτερα η αγορά εργασίας αλλά υπάρχει ένας μηχανισμός δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Ακούγεται σαν κάτι το μεγάλο για το μέλλον προφανώς, αλλά τώρα στη συζήτηση που θα γίνει για τον προπολογισμό της Ένωσης μπορούμε να εισαγάγουμε μία αλλαγή αν και γνωρίζουμε βεβαίως πως ε, ε, με 1% του ΑΕΠ της ε, Ένωσης δεν θα είναι πολύ μεγάλο ανθρωπιδικός ρόλος αλλά και από την πλευρά των εσόδων υπάρχει πλέον ένα επιχείρημα για φόρο επιχειρήσεων ευρωπαϊκό. Γιατί αν αλλάξουμε την λογική στο μέλλον κάποια στιγμή, στην πλευρά των δαπανών πρέπει να δώσουμε κάποια βάση στο ότι κάποια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ενίσχυσαν ε, τις οικονομικές τάσεις. Ε, π.χ. η Ισπανία έλαβε πάρα πολλά διαρθρωτικά ταμεία που ενίσχυσαν την ανάπτυξη. Εντάξει, βέβαια αυτή τη στιγμή δεν τίθεται το ζήτημα. Αν αλλάξουμε, λέει, τη λογική θα υπάρξει τέτοια συζήτηση. Τώρα για το πώς θα προωθήσουμε αυτές τις ευρωπαϊκές ιδέες ε, στο πολιτικό πλαίσιο και ποια είναι η κατάσταση. Για τη Γερμανία θα έλεγα πως υπάρχει μια σαφής ε, απόσταση μεταξύ της, και αντίφαση μεταξύ της θέσης για ρύθμιση όπου η Ελλάδα έχει ε, προωθήσει κάποιες ιδέες αλλά για την επιτήρηση Όσον αφορά την θέση της κυβέρνησης στο ΕΚΟΦΗΝ δεν έχει υπάρξει αλλαγή. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω πως ε, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε παρόντες, ε, να μιλάμε στο γερμανικό κοινό και τη Βουλή. Υπάρχει αυξημένο ρόλο του Γερμανικού Κοινοβουλίου, όχι μόνο λόγω τη συνθήκη Λισαβόνα, αλλά λόγω και τη απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου και νομίζω πως υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από βουλευτές, όχι μόνο από την αντιπολίτευση. Δεν είναι θέμα κυβέρνηση αντιπολίτευσης, αλλά και τα κόμματα της κυβέρνησης ασχολούνται περισσότερο με τα ευρωπαϊκά ζητήματα και κάποιοι βουλευτές είναι πιο φιλοευρωπαίοι από ότι η κυβέρνηση ίσως. Οπότε ίσως αυτό είναι ενδιαφέρον και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επόμενος γύρος, Πασκάλ Καμφά. And then και σαν Ένα λεπτό ο καθένας. Όχι, όχι, εγώ ε, με ένα λεπτό δεν βολεύομαι. Λοιπόν, Νομίζω ότι το, το, το, το, το θέμα θίγει πραγματικά την ουσία και δεν είναι από ευγένεια δηλαδή, από πεποίθηση το λέω. Μία από τις προκλήσεις της έκθεσης της Περβάνς, ε, κατά τη γνώμη μου, είναι το να δοθεί ένα περιεχόμενο στην οικονομική διαχείριση της Ευρώπης και το Κοινοβούλιο να μπορέσει να συμφωνήσει με αυτήν. Εγώ θα ήθελα να προτείνω μερικές ιδέες και να ακούσω τη γνώμη σας για αυτές. Πρώτο, η εξέλιξη της σχέσης μεταξύ μισθού και παραγωγικότητας. Αυτό το εξηγεί την υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας ή εξηγεί την υπερανταγωνιστικότητα ορισμένων χωρών έτσι όπως φαίνεται στο τρέχον ισοζύγιο. Και είναι ένα θέμα για μακροοικονομική συζήτηση. Τώρα, για το δημόσιο χρέος. Δεν έχουμε ένα κοινό εργαλείο εποπτείας. Και αν ναι, ποιο πρέπει να είναι αυτό. Περνάει μέσα από την μακροπροληπτική εποπτεία ή και από άλλα μέσα. Να ας πούμε τι έγινε με την κατάχρηση στον τομέα των, της οικοδομής, ε, των, των οικοδομών στην, στην Ισπανία. Δηλαδή τελικά εκεί το, το, το, ποσοστό ε, χρέωσης, ε, υπερχρέωσης ε, των οικοκυριών πραγματικά την άχτηκε στον αέρα μέσα από αυτήν την πολιτική κατοικία που υπήρξε. Η Board, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα μπορούσαν ίσως να προτείνουν ας πούμε στις ισπανικές τράπεζες να αυξήσουν το capital requirements για τα δάνεια στην ε, Ισπανία έστω και αν είναι μια γαλλική γερμανική τράπεζα που δίνει τα δάνεια στην Ισπανία. Τώρα για το έλλειμμα του τρέχοντος ισοζυγίου χρειάζεται ίσως ένα σύστημα σε τρία επίπεδα να έχουμε ας πούμε μία ψαλίδα όπου τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα απορρέουν από μία κανονική κατάσταση αλλά άμα ξεπεράσουν ένα κατόφλι τότε θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει πρόβλημα ή δεν υπάρχει πρόβλημα και άμα ανοίξει ακόμη παραπάνω η ψαλίδα τότε θα πρέπει να διαπιστωθεί ποιο είναι το πρόβλημα και να συζητηθεί. Και μιλάω εδώ για το ΑΕΠ ε, το οποίο συνδέεται με τον υπόλοιπο κόσμο και όχι μόνο το ισοζύγιο πληρωμών. Λοιπόν, ο κύριος Πιζανή Φερή συμφωνεί με αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλια που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Εγώ δεν είμαι από χώρα μέλος της Ευρωζώνης ο υποχρεωτικός συντονισμός των οικονομικών πολιτικών, των φορολογικών πολιτικών, ε, ο δανεισμός ε, τελευταίας καταφυγής, η ε, προσφυγή στο Διεθνές Μισματικό Ταμείο, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και συζητήθηκαν εντόνως στην Ευρωζώνη. Αλλά θα μπορούσαμε να εξετάσουμε μέσα σε λίγα λεπτά πώς αυτή η αυξημένη συνεργασία και συντονισμός στην Ευρωζώνη μπορεί να επηρεάσει τα μέλη τα οποία δεν είναι τμήμα της Ευρωζώνης. Και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Ποιος θέλει να απαντήσει στην ερώτησή σας. Διαλέξτε ένα, γιατί δεν έχουμε, το χρόνο. Εγώ θα ήθελα να ακούσω σχόλια από όλους τους ομιλητές του πάνελ. Eh, ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μα η κρίση στην Ισπανία ε, είναι ε, αποτέλεσμα διακίνησης ε, κεφαλαίων και με διασυνοριακό χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν η μακροεποπτεία είναι ουσιαστικότατη. Και εντάξει είναι σημαντικότατη η ανάπτυξη, σημαντικό στοιχείο της δημιουργίας δημοσίου χρέους, αλλά πρέπει να δούμε και το ιδιωτικό χρέος τι γίνεται. Δύο ερωτήσεις στον κύριο Πιζανή. Μίλησε για την διαφορά μεταξύ της συνυπευθυνότητας, της συνυπευθυνότητας και της ε, μη παροχής ε, βοήθειας. Αλλά αυτές τις αρχές όμως, δεν τις, αυτές οι αρχές δεν διέπουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Τι, ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν τα ευρωομόλογα σε αυτού του είδους την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Μιλήσατε επίσης για τους μισθούς πώς ε, θα μπορούσαμε να θέσουμε και, την, και την, τους μισθούς ε, μέσα σε αυτήν την μελλοντική οικονομική κατάσταση. Νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσετε εσείς ε, κύριε Βυζάνη, γιατί ο Πασκάλ, η Πασκάλ απευθύνθηκε σε εσάς και μετά θα ακούσουμε και τους άλλους δύο συναδέλφους σας. Για το θέμα του Πασκάλ Κενφά. Λοιπόν, μισθή παραγωγικότητα, βεβαίως. Μα αυτή είναι και η βάση δηλαδή για την παρακολούθηση των πραγματικών ισοτιμιών. Και σε αυτή τη βάση θα πρέπει να αρχίσουμε να φτιάχνουμε δείχτες ε, και στοιχεία κρίσης. Τώρα για το τρέχον ισοζύγιο που συνδέεται με αυτά. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ να υπάρχει ένα κατόφλι συναγερμού. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε κατόφλια ε, του ίδιου τύπου με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Αλλά όμως μπορούμε να πούμε ότι από ένα κατόφλι και μετά ξεκινούμε μια εξεταστική διαδικασία. Και αυτή θα μπορούσε να είναι η έκθεση που θα πρέπει να συντάξει η Κομισιόν για να πει αν η κατάσταση του τρέχοντος ισοζυγίου των ε, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δημιουργεί πρόβλημα ή όχι. Υπό τον όρο όμως ότι δεχόμαστε ανοιχτά ότι μπορούμε να έχουμε και τις δύο απαντήσεις. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε απαντήσεις που λένε όχι, έχουμε ένα σημαντικό έλλειμμα, αλλά αυτό είναι το έλλειμμα ή αλλιώς να, πούμε, να έχουμε και την αντίθετη απάντηση. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Δεν χρειάζεται εδώ να μολύνουμε τη λογική του Συμφώνου Σταθερότητας, είναι εντελώς διαφορετική λογική. Για το ιδιωτικό χρέος Μα <coughs> η δυσκολία είναι η ευθύνη της χώρας υποδοχής, η κατάσταση των τραπεζών και η ευθύνη της χώρας προέλευσης. Όταν όλα αυτά συμπίπτουν, μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα της οικονομικής σταθερότητας σε μια χώρα από τις, ε, εξετάζοντας τις τράπεζές τους. Αλλά όταν έχουμε, είμαστε σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα κάτι τέτοιο δεν λειτουργεί. Χρειάζεται λοιπόν από την αρχή να δεχτούμε το ότι δουλεύουμε μέσα σε ένα σύστημα ολοκληρωμένο και να πούμε ότι ο έλεγχος των τραπεζών δεν είναι καλή λύση. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να βασιζόμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι ενδιάμεση κατάσταση και η οποία δεν θα ισχύει αύριο. Ε, όταν δηλαδή οι περισσότερες χώρες της κεντρικής Ευρώπης θα έχουν μπει στην Ευρωζώνη. Τώρα για τους ε, μισθούς ε, ναι, απάντησα και απαντώντας τον κύριο Κεμφά. Τώρα για το θέμα της, ε, ε, της ε, μη παροχής βοήθειας και της ε, αρρωγής, μα αυτό είναι κάτι αυτονόητο. Διότι οι συνθήκες είναι σαφέστατες, έχουμε τον κοινοτικό προϋπολογισμό είτε αναλαμβάνονται λαμβάνονται διμερώς ευθύνε είτε κοινοτικά. Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν νομικά η κατάσταση δεν είναι ακριβώς η ίδια για την αρχή, την ίδια, δεν υπάρχει λόγος να πούμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά τη βοήθεια σε ένα κράτος ή τη διαφορά σε δύο κράτη. Μα δεν υπάρχει καμία διαφορά. Είναι ίσως νομικό το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά το ερώτημα για το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο το, το αντιλαμβάνομαι. Εγώ είχα ασκήσει κριτική στα τελευταία χρόνια την απροθυμία ορισμένων κρατών μελών και της Γερμανίας να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της Ευρωζώνης ως τέτοια. Βλέπω πως υπάρχει μια ανησυχία για ένα πιθανό χάσμα. Βεβαίω θα είναι θεσμικό εάν ε, διευρυνθεί η Ευρωζώνη, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό αποκλεί πολιτικούς στενότερους δεσμούς με τις χώρες που αυτή τη στιγμή δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης. Οι δε θεσμικοί δεσμοί θα είναι πάντα ισχυροί και είναι κάτι το απαραίτητο εάν ε, θεσμοποιηθεί η Ευρωζώνη εντό Ένωση να παραμείνουν αυτοί οι δεσμοί. Π.χ. όπω υπάρχει μεταξύ Eurogroup και Εγκοφίν, καθώ συνεδριάζουν την προηγούμενη μέρα και μετά η συζήτηση μεταφέρεται στου 27 υπουργού. Κάτι ανάλογο μπορούσε να γίνει και στο Ιαρινό Συμβούλιο, όπου μιλάμε για οικονομική πολιτική ανταγωνιστικότητα και θα μπορούσε πρώτα απ' όλα να γίνει μια μικρή συζήτηση, η οποία μετά θα μπορούσε να μεταφερθεί στις 27. Οπότε πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να μας εμποδίσει να σκεφτούμε στα προβλήματα τη ΟΝΕ τέτοια εσωτερικά. Τώρα για το θέμα των μισθών. Για να προσθέσω κάτι σε αυτό το οποίο είπα πριν για την ενίσχυση της Ευρωζώνης, ο μακροοικονομικός διάλογος είναι κάτι που δεν έχει αξιοποιηθεί η λεγόμενη διαδικασία της κολονίας του 1999 και εδώ πέρα πρέπει να δούμε το εάν μπορούν να εμπλακούν οι κοινωνικοί εταίροι σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά όταν μιλάμε για ανταγωνιστικότητα μιλάμε για μισθούς και έχουμε την εξή κατάσταση. Η κυβέρνηση μπορεί σε πολύ μικρό βαθμό μόνο να επηρεάσει το τι κάνουν στις διαπραγματεύσεις εταίροι της. Σύντομα, Νομίζω πως η δημιουργία του ευρώ είναι μακράν η πιο προχωρημένη μορφή ολοκλήρωσης που είχαμε ποτέ και αυτό έχει συνέπειες για την οικονομική διακυβέρνηση και ε, ποσοτικά και ποιοτικά διαφορετικές από τις ε, απαιτήσεις από το υπόλοιπο κοινοτικό και εκτιμένο. Και αυτό άρα αναπόφευκτα έχει συνέπειες για αυτούς που είναι μέσα και για αυτούς που είναι έξω. Αυτό το οποίο είναι κρίσιμο είναι πως πρέπει να κρατήσουμε όλη την πόρτα ανοιχτή και τους δεσμούς μεταξύ των μέσα και των έξω, ώστε να τον πιο στενό σε ένα τελευταίο σημείο. Ανέφερα τις ε, φορολογικές πολιτικές και νομίζω τις αναφέρατε και εσείς. Εγώ υποθέτω και ελπίζω πως οι φορολογικές ε, πολιτικές θα τονιστούν περισσότερο, όχι μόνο για τα μέλη της Ευρωζώνης αλλά και για τους 27. Οι δύο τελευταίοι, ο Ατμαρκάρας και Περβάμς Μπερές. Ναι, κυρίες μου και κύριοι, αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει είναι ότι είμαστε μια πολύ γενική συζήτηση και μιλάμε για διακυβέρνηση. Το ερώτημά μου προς σας είναι Μήπως δεν είναι ένα από τα προβλήματά μας το ότι δεν τηρούμε τους κανόνες που ήδη έχουμε σε πολλές περιπτώσεις. Είναι απολύτως απαραίτητο να μιλάμε για νέες μεθόδους διακυβέρνησης. Μήπως είναι σημαντικό πρώτα να πούμε ποιες μεθόδους διακυβέρνησης έχουμε τώρα και τι μπορούμε να κάνουμε για να τις στηρίσουμε αυτές. Δεν ξεκίνησαν όλα με την κρίση. Πολλά ξεκίνησαν με την μη τήρηση των κανόνων μας. Κατ' η κρίση. Και δεν ισχύει το ότι όλα όσα έχουμε είναι άσχημα ή ότι δεν είχαμε τίποτα. Ήμασταν σε καλό δρόμο μέχρι την κρίση. Έχουμε λίγα ίσως και το θέμα είναι πού χρειαζόμαστε συμπληρωματικά μέτρα γιατί αυτά τα οποία έχουμε δεν επαρκούν. Αυτό είναι το αποφασιστικό ερώτημα για μένα. Εγώ έχω μία ερώτηση, μία, μία συγκεκριμένη ερώτηση για τον ε, κύριο Φερή. Είπατε ότι σε εθνικό επίπεδο πρέπει να αναπτύξουμε τα εθνικά μας μέσα για να ασχοληθούμε με την ανταγωνιστικότητα ε, και να δούμε και το ζήτημα των μισθών. Μήπως μπορείτε να μου το αναλύσετε τώρα για τα φορολογικά. Μα φυσικά συμφωνώ, αλλά ανησυχώ όμως ιδιαίτερα. Διότι ακούσαμε τις προάλλες τον Μάριο Μόντι να μας λέει τι σκέφτεται και τι έχει κατά νου ως προς την εντολή που έχει αναλάβει και αισθάνθηκα ότι υπήρχε μια προδοσία τουλάχιστον ως προς το αρχικό πακέτο. Η εντύπωση που είχαμε προηγουμένως ήταν ότι το θέμα της ολοκλήρωσης εσωτερικής αγοράς ήταν ένα σημείο πολύ σημαντικό για την ημερήσια διάταξη αλλά ε, όσον αφορά στο, ε, στο φορολογικό πραγματικά η στόχη είναι χαμηλή. Και άμα δω και το έγγραφο 2020, σε τεμπέ γράφει, δηλαδή πάση τε, μη αναφερόμενο. Λοιπόν, είναι τόσο επίγον το θέμα που πλάθ εξαφανίστηκε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε λοιπόν στο τέλος άμα προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Και πραγματικά εγώ συχαίνομαι πια, δεν αντέχω άλλο, έχω σκάσει με τη θεσμική συζήτηση. Αλλά υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Λέμε ότι δεν θέλουμε κυβέρνηση δικαστών. Ναι, αλλά τι κάνουμε, φτιάχνουμε μια κυβέρνηση κεντρικών τραπεζικτών. Και αυτό πάλι δεν πάει καλά. Όταν λέτε εσείς ότι το θέμα της διάρθρωσης μεταξύ μακροοικονομίας και μακροληπτικής εποπτείας κλπ είναι κάτι ε, πραγματικά πολύ σημαντικό, δηλαδή μακροληπτική εποπτεία, μακροοικονομική παρακολούθηση. Αλλά πραγματικά πώς θα καταφέραμε να βρισκόμαστε σε, μια, σε τέτοιο χάος όπου, όπου τελικά τι γίνεται πάνω στην ελληνική κρίση που αυτό που έπρεπε να συγκληθεί θα ήταν μια διάσκεψη κορυφής ευρώ, ο Ζαπατέρο δεν την καλεί. Γιατί, γιατί ο κύριος Βαν Ρομπόη δεν ξέρω τι και υπήρχε ανταγωνισμό σε θεσμικό επίπεδο. Ο κύριος Όλι Ρεν δεν τα καταφέρνει, ο κύριος Γιούνκερ δεν τα καταφέρνει και η κυρία Σελγάδο ούτε. Απολύ εκνευρίζομαι, αλλά είναι εντελώς άχρηστο γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα συμφωνήσουμε. Αλλά τέλος πάντων πραγματικά. Πραγματικά, πραγματικά, δηλαδή πραγματικά βαρεθήκαμε να λέμε έχουμε όλα αυτά τα μέσα, όλα αυτά τα μέσα και, και να μην φτιάχνουμε τίποτα. Πρέπει να ξεπεράσουμε την ανικανότητα των κρατών μελών και έχουμε τις ευθύνες μας για αυτά. Και πρέπει και εμείς να τα βρούμε για το τι θα προτείνουμε δηλαδή. Ευχαριστώ προς τον κύριο Καράς. Συμφωνώ πλήρως για την Ελλάδα μαζί σας. Αλλά ποιοι είναι οι κανόνες που δεν σεβάστηκε η Ισπανία. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει Η Ισπανία ήταν νομότυπη, σεβάστηκε τους κανόνες. Ε, είχε δημοσιονομικό έλλειμμα. Φυσικά δεν βάζω και τις δύο χώρες στο ίδιο καλάθι. Φυσικά υπάρχει πρόβλημα στην Ισπανία παρότι δεν είναι το ίδιο με το πρόβλημα της Ελλάδας. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι η Ισπανία παρακολούθησε και σεβάστηκε και τήρησε όλους τους κανόνες. Όχι, δεν συμφωνείτε. Ένα από του λόγου που έχουμε πρόβλημα είναι ότι κανένα δεν σεβάστηκε τη στρατηγική τη Λισαβόνα. Κανένα. Εφόσον κανένα δεν την σεβάστηκε, τότε δεν υπάρχει διαφορά. Είμαστε ισότιμε προ αυτό. Η Γερμανία Η Γερμανία δεν τη σεβάστηκε. Συμφωνώ ότι το τμήμα του προβλήματος είναι το θέμα της εφαρμογής. Αλλά τμήμα του προβλήματος. Και υπάρχει κι άλλο πρόβλημα. Και το γεγονό ε, ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα για την εφαρμογή. Ισχύει και αντίστροφα αυτό. Τα μέσα ανταγωνιστικότητες. πραγματικά ορισμένες χώρες παρακολουθούν την ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή όταν μπήκανε στη Ζενευροζώνη ε, έκαναν σημαντικό έργο για να βρούνε τι μέσα θα βρούνε για να αποφύγουν σημαντικές ανσημετρίες. Η Φιλανδία έκανε πολλή δουλειά. Άλλες χώρες όμως δεν το κάνανε, είπαν εντάξει μπήκαμε στο ευρώ και ωραία, τελειώσαμε. Και ανέθεσαν αυτή τη δουλειά στις ε, τράπεζες κλπ. Αυτή η δουλειά λοιπόν πρέπει να γίνει τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι το μέσο είναι το ίδιο, εξαρτάται και από τη διάρθρωση των διαπραγματεύσεων, αν έχουμε χώρε με κεντρική διαπραγμάτευση, με αποκεντρωμένη διαπραγμάτευση, είναι πιο εύκολο για τι χώρε με συγκεντρωτική διαπραγμάτευση. Πέρα δηλαδή από το γεγονός ότι χρειάζεται και πολιτική παρακολούθηση. Τώρα η ερώτηση είναι περισσότερο του Λουκά βέβαια. Για τις κεντρικές τράπεζες ε, και για το κατά πόσο πρέπει να διατάζουν. Μα αυτό δεν είναι καν ευκταίο για τους ίδιους ε, τους ε, κεντρικούς τραπεζίτες. Δηλαδή δεν είναι ευκταίο η μόνη αρχή η οποία να έχει πραγματική αποτελεσματικότητα να είναι η κεντρική τράπεζα. Και να έχουμε αυτή την κεντρική τράπεζα με συνεχώς διευρυμένες αρμοδιότητες που θα οδηγήσει σε μία αντίφαση μεταξύ της εντολής της και των πραγματικών της αρμοδιοτήτων. Είναι αλήθεια ότι έχουμε κανόνες οι οποίοι δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά. Η συμφωνία, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης έγινε όλο και πιο χαλαρό, ευέλικτο για να το πω α, έτσι, μαλακά, ε, υπήρχαν ένοχοι πολύ πριν εμφανιστούν στη σκηνή οι Έλληνες. Επίσης, είναι αλήθεια, δεν έχουμε και σε άλλους τομείς κανόνε. κανόνες. Παραδείγματο χάρη ρύθμιση και κανόνες. Κατά την άποψή μου, η πρόσφατη κρίση εξέθεσε όχι μόνο το πρόβλημα της ανεπάρκειας των κανόνων, αλλά το βαθμό σύγχυσης και το βαθμό άρνησης α, μέσα στον οποίο ζει και κινείται η πολιτική μας, η, ζουν και κινούνται οι πολιτικοί μας ηθήνοντες. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ύπαρξη, η, η ανεπάρκεια ή η ανυπαρξία κανόνων. Είναι πολύ πιο ουσιώδες θέμα. Έχετε την τελευταία λέξη. Συμφωνώ με αυτό το είπε ο κύριο Κάρα, Είναι και θέμα και διαδικασίας. Και... Αλλά και δικτών. Στην παραδοσίασή μου προσπάθησα να δείξω γιατί δεν λειτουργήσε η εφαρμογή. Δεν το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Εκτός και αν υπάρξει μεγαλύτερη μεταφορά αρμοδιοτήτων. Και αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Θα πρέπει λοιπόν να δημοσιοποιήσουμε το θέμα, να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση του κοινού ε, και αυτό μας το δείχνει και η ελληνική κρίση. Υπάρχουν και άλλες κρίσεις που ελοχεύουν, της Ισπανίας κτλ. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι και η γερμανική συζήτηση αλλάζει σε σχέση με το μοντέλο ανάπτυξης. Ε, και στο εσωτερικό, πέρα από τους ξένους, έτσι, αρχίζει να γίνεται μια κοινοβουλευτική συζήτηση για το μοντέλο ανάπτυξής μας στη Γερμανία. Κάτι αλλάζει, σιγά σιγά. Και για τους λόγους που σας εξήγησα, συμφωνώ ότι τα πράγματα δεν είναι επαρκή, δεν είναι ικανοποιητικά. Αλλά ρεαλιστικά, αν το δούμε, ο μόνο τρόπο που μπορούμε να προχωρήσουμε ε, είναι αυτή η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελείωσε το πρώτο πάνελ. Σα ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσής μας. Έχουμε άλλους τρεις εξαίρετους ομιλητές. Τα βιογραφικά τα έχετε, δεν θα πω πολλά. Πέντρο Πέρες πρώτα απ' όλα, μετά από πολλά χρόνια στην διοίκηση ε, είναι τώρα πρόεδρος ε, σε κάποια εταιρεία μετά έχουμε την κυρία Αν Πέτιφορ που έγινε γνωστή μέσω του ότι το 2000 ξεκίνησε το έργο Jubilee 2000, μια καμπάνια για να βοηθούν οι φτωχότεροι των φτωχών ε, χωρών για να απαλλαγούν από τα χρέη τους πολλών δισεκατομμυρίων που αποτέλεσε παράδειγμα πολλών άλλων παρόμοιων πρωτοβουλίων και τέλος έχουμε τον Ιταλό συνάδελφο, τον κύριο Λούκα Παουλάτσι, επικεφαλής οικονομολόγο του Συνδέσμου Βιομηχάνων της Ιταλίας. Απόφυτος ε, οικονομικών του Πανεπιστημίου Μποκόνη. Οπότε σας καλωσορίζω. Ε, κύριε Πέρες. Μπορείτε να μιλήσετε και ισπανικά, ό,τι γλώσσα επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ έλεγα κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετέχω σε αυτήν την Επιτροπή που εξετάζει θέματα πάρα πολύ σημαντικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της. Θα ήθελα καταρχήν να τονίσω το εξή ότι με τις συζητήσεις που κάνουμε, με ό,τι βλέπουμε στη... και διαβάζουμε στα ΜΜΕ, φαινότανε ότι η κρίση επήλθε και οξύνθηκε διότι υπήρχε κακή φορολογική διαχείριση. Και αποκρισταλώθηκε η άποψη ότι η κρίση οφείλεται σε μία ανεπαρκή και ακατάλληλη εναρμόνιση της φορολογικής πολιτικής και της ακαταλληλότητας επίσης των μέτρων που δεν ελήφθηκαν έγκαιρα. Υπάρχει ένα άρθρο σχετικά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πως το όλο νομισματικό πρόβλημα είναι αυτό που οδήγησε στην κρίση. Λοιπόν, την νομισματική πολιτική κατά συνέπεια θα πρέπει να την δούμε ευρύτατα. Όχι απλώς ιδέοντας επιτόκιο με πληθωρισμό. Να δούμε πώς έχουμε τις διάφορες διακυμάνσεις των νομισματικών ροών και των αγορών για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα που κατά τη γνώμη μου είναι εμφανές. Σήμερα η Κεντρική Τράπεζα η οποία εισήγαγε εξαιρετικούς μηχανισμούς για να εξετάσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση τόσο των οικογενειών όσο και των οικογενειών δεδομένου ότι οι αγορές έχουν ε, καταρρεύσει. Πώς διαρθρώθηκαν λοιπόν τα μέτρα. Πώς δηλαδή θα επανέλθουμε σε παλιούς μηχανισμούς ε, για την δανειοληψία δεδομένου ότι δεν υπήρχε δυνατότητα, πιστοληπτική δυνατότητα στην Ευρώπη. Οι τράπεζες λοιπόν ξεκίνησαν με αυτούς τους έκτακτους και εποχιακούς μηχανισμούς Λοιπόν, η φορολογική πολιτική λοιπόν μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία κινήτρων για τον παραγωγικό μηχανισμό και να αντισταθμίσει την έλλειψη ρευστότητας και να δημιουργήσει νέα δραστηριότητα αλλά η φορολογική πολιτική δεν μπορεί να υποκαθιστά συνεχώς την έλλειψη μιας σωστής νομισματικής πολιτικής. Για να το πω με άλλα λόγια, εάν με την τραπεζική ρύθμιση και την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας και όταν λέω εγώ τραπεζική ρύθμιση εννοώ ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας της αγοράς και του τραπεζικού συστήματος ούτως ώστε το ρευστό να μπορεί να πηγαίνει προς τις επιχειρήσεις και προς τις οικογένειες. Βέβαια, για να γίνει κάτι τέτοιο η φορολογική πολιτική έχει περιορισμένες δυνατότητες και έχει φτάσει πλέον στα όρια. Και αυτή η ανησυχία εκφράστηκε και στις συζητήσεις που είχαμε σήμερα το πρωί. Θέλω λοιπόν να επιμείνω λέγοντας ότι η χρηματοδότηση του παραγωγικού μηχανισμού είναι κάτι το κατεπήγον δεν μπορούμε εμείς να εξαντλήσουμε τα περιθώρια της φορολογικής πολιτικής και να περιμένουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε αναζωγόνηση της οικονομικής δραστηριότητας. Και για να επανέλθω στα φορολογικά. Ως συνέπεια αυτής της εμπειρίας, εμείς αντλήσαμε διδάγματα ώστε στο μέλλον να είμαστε πιο προσεκτικοί για τη δημιουργία ενός φορολογικού χώρου και όταν μιλάω εγώ για χώρο μιλάω για φορολογική ικανότητα η οποία να επιτρέπει στις κυβερνήσεις να διαχειρίζονται πιο ευέλικτα την κατάσταση. Αυτό όμως είναι μελλοντολογία. Σήμερα η ανησυχία μας θα πρέπει να επικεντρώνονται στο η μείωση του δημοσίου ελλείμματος να γίνει κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ζημιές για τον παραγωγικό μηχανισμό. Είναι λοιπόν όλα αυτά πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε δηλαδή να διασώσουμε τις επενδύσεις, τις υποδομές, στην παιδεία, στην έρευνα, ούτω ώστε δηλαδή όλες αυτές τις δαπάνες, ούτω ώστε η, η Ευρώπη μετά από την κρίση να βγει ενισχυμένη. Αδιαμφισβήτητα η κρίση και αναφέρθηκε πολλές φορές σήμερα το πρωί, η κρίση λοιπόν απέδειξε ότι θεσμικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν καλά προετοιμασμένη. Σίγουρα στην συνθήκη της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ρίχθηκε ο σπόρος για να αναπτυχθεί η ναι μέσα στο χρόνο. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η στιγμή κατά την οποία ασκείται η κριτική μιας οικονομικής πολιτικής ή μιας φορολογικής δράσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Έτσι λοιπόν Ούτε η Κεντρική Τράπεζα, ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε και οι Κομισιόν ήταν έτοιμες, είχαν μια γρήγορη αντίδραση. Αυτό είναι ένα δίδαγμα και που θα πρέπει να το θυμόμαστε στις μελλοντικές μας λήψεις θέσεων. Επίσης, όπως είπαν και άλλοι, η έξοδος από αυτήν την κατάσταση χρειάζεται ε, μία εμβάθυνση στο πώς θα δημιουργήσουμε περισσότερη ένωση στην Ευρώπη. Περισσότερη ένωση μέσα από μια καλύτερη και πιο εναρμονισμένη δημοσιονομική ρύθμιση. Εδώ αυτό γίνεται, αλλά από ό,τι λένε, αλλά εμείς από τον ιδιωτικό τομέα το βλέπουμε να ολοκληρώνεται πολύ αργά διότι είναι τρία χρόνια που ξεκίνησε η κρίση και ακόμη εμείς συζητάμε βασικά ε, και στοιχειώδη θέματα νομισματικής ε, διαχείρισης και θέματα ρύθμισης της κρίσης. Δεν χρειάζεται να τροποποιήσουμε το στόχο της Κεντρικής Τράπεζας διότι έτσι όπως ορίζεται από τη συνθήκη είναι να εστιάζει τη δράση του ε, εγγυόμενο τη σταθερότητα αλλά όταν έχει εγγυηθεί πια τη σταθερότητα θα πρέπει να εστιάζει την ανησυχία του στην εξυπηρέτηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι φανερό σήμερα, έχουμε σταθερότητα των τιμών. Και η σταθερότητα των τιμών βραχυπρόθεσμα δεν απειλείται. Αλλά όμως εμείς τη βλέπουμε η Κεντρική Τράπεζα ανησυχεί περισσότερο για την απόσυρση των εκτάκτων μηχανισμών πριν αρχίσει δηλαδή να προχωρεί θετικά η πιστοληπτική ικανότητα μέσα στην Ένωση. Χωρίς δηλαδή να εξυπηρετούνται οι στόχοι για τη δημιουργία ανάπτυξης και πώς εμείς θα μιλήσουμε για συντονισμό των φορολογικών πολιτικών όταν ο προϋπολογισμός της Ένωσης είναι ελάχιστος και οι ε, δυνατότητες που έχει αυτός ο προϋπολογισμός είναι σχεδόν γελίες αν μου επιτρέπετε φυσικά την έκφραση συζητείται σήμερα η φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών πράξεων αλλά αυτή όμως η φορολόγηση πρέπει να είναι παγκόσμια πέρα δηλαδή από τον φόρο αυτό να τον πληρώνουμε μόνο στην Ένεση και στην Αποανατολή πρέπει να πληρώνεται και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πρέπει λοιπόν εμείς να ρυθμιστούμε και να διορθωθούμε μέσα στην Ένωση. Και από εκεί θα, βρει, θα αντλούσαμε και τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερους προ, πόρους για μεγαλύτερα προγράμματα δαπανών. Να έχει επίσης η Ένωση και γρήγορα μέσα παρακολούθησης για να μπορεί δηλαδή να παρακολουθεί και το τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Ε, θέλω να μιλήσω για την ε, νέα πράσινη συμφωνία, Green New Deal. Ε, στην τελευταία συνεδρίαση είπαμε ότι δεν πρέπει να επανέλθουμε στα ίδια τα συνηθισμένα. Είναι πολύ αργά. Όχι απλώς επανήλθαμε, αλλά ο τραπεζικός τομέας ε, επανήλθε στα ίδια τα συνηθισμένα επαυξημένα. Έχουμε μια κατάσταση τώρα όπου ένα τρίτο του ΑΕΠ της ε, Eurozone, μιλάμε για δημόσιο χρήμα, πηγαίνει για την υποστήριξη των τραπεζών. Του έδωσε τη δυνατότητα οι τράπεζε έτσι να ανακάμψουν πολύ γρήγορα και να ξαναρχίσουν. Οι χρηματαγορές ανθούν, τα μπόνους. Αλλά έχουμε ε, και επαγιοποίηση του τραπεζικού τομέα. Φύγαν οι ανταγωνιστές. Νομίζω ότι το business ε, τα πάει μια χαρά, ας πούμε είναι όπως πριν και καλύτερα. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα, ξεκινώντας, να πω ότι υπάρχουν κάποια βασικά λάθη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα οικονομικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την ανάκαμψη. Και ένα από αυτά μας το ανέφερε ο, ο καθηγητής Χάλομπερκ στο έγγραφό του. Είπε ότι οι αγορές δίνουν τα χρήματα που χρειάζονται τα κράτη για να χρηματοδοτήσουν το χρέος του. Θέλω να το αμφισβητήσω. Θέλω να πω ότι οι κεντρικές τράπεζες και είναι η, η, πηγή από την οποία προέρχονται τα χρήματα. Δημιουργούν ε, χρήματα, πίστη και το κάνουμε στη χώρα μου από το 1694. Τότε δεν το λέγαμε quantitative easing, αλλά επιχειρήσεις στην ανοιχτή αγορά. Από το, το 2009 η ΕΚΤ δημιούργησε 442 δισεκατομμύρια για τις αγορές και συμμετείχαν 1.192 ε, τράπεζες σε αυτό το σύστημα ε, ενισχυμένης ε, πιστοτικής στήριξης. Στη χώρα μου και στις ΗΠΑ, τα δύο τρίτα του ΑΕΠ πήγαν σε αυτού του είδους τη στήριξη. Στη Βρετανία η Τράπεζα της Αγγλίας έμεσα μέσω των αγορών χρηματοδοτεί το κυβερνητικό χρέο. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Θα πρέπει πραγματικά να το συνειδητοποιήσουμε. Ε, ο Κέιν προσπάθησε να το εξηγήσει στη δεκαετία του 30 στου οικονομολόγους και δεν το κατάλαβαν. Θα πρέπει να το καταλάβουμε όμω εμείς σήμερα. Η, πέρυσι η Τράπεζα τη Αγγλίας δημιούργησε από τίποτα 200 δισεκατομμύρια στερλίνε για αυτό το quantitative easing τα έδωσε στις αγορές μέσω κυβερνητικών ομολόγων και άλλων τίτλων και οι, τα αγόρασαν οι τράπεζες. Αυτό βοήθησε για να χρηματοδοτήσουμε το κυβερνητικό έλλειμμα της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά είναι ουσιαστικά πράγματα. Πρέπει να τα καταλάβουμε. Και αν δεν τα καταλάβουμε, δεν θα καταλάβουμε καθόλου την πίστη, το χρήμα, πώς λειτουργεί και κυρίως το τραπεζικό χρήμα. Δεν είναι κατανοητό από τους οικονομολόγους. Ο Κέις προσπάθησε να το εξηγήσει. Και άλλοι οικονομολόγοι προσπάθησαν να το εξηγήσουν. Αλλά οι μοντέρνοι οικονομολόγοι, οι σύγχρονοι οικονομολόγοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Ε, δηλαδή, το τραπεζικό χρήμα δεν είναι αγαθό. Δεν υπόκειται στους κανόνες προσφορά και ζήτηση. Δεν είναι όπως ε, το πετρέλαιο, το, ο χρυσός ή του λίπε. Είναι απεριόριστο στη, σε όγκο και πρόσφατα είδαμε όταν ο κύριος Μπερνάνκε ε, στην τηλεόραση σε μια πρώτη συνέντευξη που έδωσε ένας διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος πού βρήκε 160 δισεκατομμύρια δολάρια να πληρώσει στην AIG που δεν είναι τράπεζα. Είναι, ήταν μάλλον, μια ασφαλιστική εταιρεία. Αλλά λόγω της κρίσης ε, δόθηκε ένας λογαριασμός ε, στη Fed Και όταν του είπαν, πού βρήκατε αυτά 160 δις, είπαν, χρησιμοποίησαμε απλώς το κομπιούτερ για να βάλουμε το νούμερο του λογαριασμού που έχει στη Fed Και 160 δισεκατομμύρια εμφανίστηκαν εν μία νυχτή. Ευτυχώ, γιατί αν δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, λέω εγώ, τότε θα είχαμε μια πιο βαθιά κρίση. Ε, το παράπονο μου είναι ότι δόθηκε χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Επομένως, ε, το πρόβλημα της καθεστικίας άποψης είναι ότι πρέπει να έχουμε αποταμιεύσεις στην τράπεζα για να δημιουργηθεί οικονομική δραστηριότητα. Η Ελλάδα θα πρέπει να συσσωρεύσει αποταμίευση στην τράπεζά της για να δημιουργήσει οικονομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει εισόδημα για να πληρώσει το τεράστιο ιδιωτικό χρέος που υπάρχει στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρωζώνη, από τη μία και από την άλλη το δημόσιο χρέος που έχει σωρευτεί. Αν παρακολουθήσετε τη λογική ότι καταρχάς πρέπει να δημιουργήσουμε την αποταμίευση για να υπάρξει οικονομική δραστηριότητα, τότε τελικά δεν θα υπάρξει ποτέ εισόδημα. Και αυτό που εξυπακούεται είναι ότι η οικονομική δραστηριότητα περιορίζεται από την αποταμίευση. Ο Keynes το συνέλαβε αυτό με φοβερή διορατικότητα. Ο... Ότι μπορούμε ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις τράπεζες ε, να μας δώσουν τα λεφτά. Ε, μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε λόγω της ε, μαγικής λειτουργίας της πίστης, της πίστοσης. Το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε της μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη, εκατομμύρια ανέργων χιλιάδες εργοστάσια, εταιρείε, ε, επιχειρήσεις που χρεοκοπούν καθημερινά, αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της δημιουργίας πίστοσης, που θα πρέπει φυσικά να την χάνει κάποια διαχείριση, να υπάρχει διαχείριση σε ένα περιβάλλον κλήρους οικονομικής δραστηριότητα. Ε, ε, μάλλον σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι πληθωριστική, όπου η υπερβολική πίστη οδήγησε σε πληθωρισμό. Και οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν το είδαν αυτό σε αυτή τη δημιουργία της πίστοσης και στη δημιουργία τίτλων μέχρι να σπάσει φούσκα. Επομένως, δεν μπορούμε να έχουμε υπερβολικά πολύ πίστη όταν υπάρχει μεγάλη οικονομική δραστηριότητα. Αλλά όταν υπάρχει έλλειψη οικονομικής δραστηριότητας, τότε θα πρέπει να δώσουμε πίστοση στο σύστημα για να δημιουργήσουμε αυτή την οικονομική κρίση για το οποίο είπε ο κύριος Περέζ. Το κάναμε. Το 1 τρίτο της, του ΑΕΠ της Ευρωζώνης μπήκε εκεί. Αλλά δεν πέρασε στους παραγωγικούς φορείς, στις εταιρείες που δημιουργούν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα και που θα δημιουργήσουν και το εισόδημα που θα πληρώσει το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος. Ένα, μια άλλη λανθασμένη προσέγγιση ε, του χρέους της Ελλάδας είναι ότι το χρέος μπορεί να αποπληρωθεί με ψηλότερους φόρους από τη μία ή από τη μείωση των δημοσίων δαπανών από την άλλη με ένα κλασικό βρετανικό τρόπο, εγώ θα πω ότι υπάρχει και τρίτος δρόμος για να πληρώσουμε το χρέος ε, μέσω της δημιουργίας εισοδήματος και είναι μάλιστα ο μόνος τρόπος, μέσω της γέννησης εισοδήματος. Αν κάνουμε α, οικονομική αφέμαξη, αν ο ασθενής δεν φάει τίποτα, ε, αποδυναμωθεί εντελώς, τότε δεν μπορεί να συμμετάσχει στην οικονομική δραστηριότητα τότε θα μειώσουμε και το δημόσιο και το ε, ιδιωτικό εισόδημα. Ένας τρίτος τρόπος για να δημιουργηθεί εισόδημα είναι μέσω των δημοσίων δαπανών. Οι δαπάνε σε δημόσια έργα. Παραδείγματο χάρη, ξοδεύουμε χρήματα ε, για να γλιτώσουμε τι τράπεζε. Ε, Χωρί όρου. Αυτό δεν είναι επενδύσει. Ξοδεύουμε έτσι τι δημόσιε δαπάνε. Αλλά αν κάνουμε, παραδείγματο χάρη, δημόσιε δαπάνε σε δημόσια έργα, περίπου, παραδείγματο χάρη στι ε, περιβαλλοντικέ προκλήσει που αντιμετωπίζουμε στο εγγύηση μέλλον. Και αυτό χρειάζεται υψηλό βαθμό θέσεων απασχόληση. Έτσι, δημιουργούμε θέσει απασχόληση, δημιουργούμε φορολογικό, φορολογικά έσοδα και νέε αποζημιώσει και αποταμιεύσει. Ε, υπάρχει ο βαθμό, εδώ το φαινόμενο του πολλαπλασιαστή, το χρησιμοποιούσε ο Κέινς. Το ξέχασαν όμως οι οικονομολόγοι, δεν, δεν χρησιμοποιούν αυτή την έννοια πλέον. Αν πει ε, σε κάποιον ότι στην Ελλάδα, πούμε, ότι πρέπει να μονώσει το σπίτι σου, πληρώνεις, πληρώνεις τους φόρους σου, εσύ πληρώνεις για αυτή τη δουλειά, ο, αυτός που κάνει την εργασία πληρώνει τους φόρους του κτλ. Αν δεν το κάνουμε αυτό, η Ευρωζώνη θα συρρυκνωθεί περισσότερο. το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και η Γερμανία είναι προκειμένου, είναι ότι αυτό το χρέος, το αποπληθωριστικό, θα διωγγωθεί όπως έγινε στην Ιαπωνία. Και θα ήθελα να σας πενθυμίσω, αγαπητοί βουλευτές, ότι η Ιαπωνία είχε ένα τεράστιο εξαγωγικό πλεόνασμα, όπως η Γερμανία. Και όμως αυτό δεν την εμπόδισε από το να βουτήξει σε, αυτή, σε αυτόν τον κικαιώνα του αποπληθωριστικού χρέους με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε την οικονομική. Αν, μειώσουμε την οικονομική δραστηριότητα και εμεί θα αντιμετωπίσουμε αυτό το, το φάσμα. Θα ήθελα να σας, δώσω, να σας δείξω αυτό το ιστορικό γράφημα. Ξεκινάει από το 1880. Ε, είναι για τα βρετανικά οικονομικά πράγματα. Σας δείχνει ότι το 1933 το έλλειμμα του δημοσίου χρέους ε, αυξήθηκε πάρα πολύ. Ο Κέινς τότε ε, έλεγξε την ε, Τράπεζα της Αγγλίας και το Βρετανικό Κορβανά και προώθησε νέες νομισματικές πολιτικές και διαχείριση και το χρέος μειώθηκε μέχρι τον πόλεμο. Η Βρετανία έπρεπε μετά να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους, περισσότερα κονδύλια, δανείστηκε περισσότερο από ό,τι είχε δανειστεί ποτέ στην ιστορία της, ε, με πολύ χαμηλά ε, επιτόκια, χάρη στον Γκέινς και στην νομισματική του πολιτική και το 1946 το χρέος μας ήταν 256% του ΑΕΠ μας τεράστιο χρέος και τα σημερινά χρέη σε αντιδιαστόλη φαίνονται γελία. Και τι έκανε μετά, άρχισε να ξοδεύει η Βρετανική κυβέρνηση. Δημιουργήσαμε τον ε, τομέα της υγείας, ε, δημόσιες, ε, δημόσιες κατοικίες, εργατικές κατοικίες, εκπαίδευση κτλ. Τι έγινε, να, έπεσε το κυβερνητικό χρέος, το κρατικό χρέος. αργά αλλά σταθερά, καθώς ανέκαμψε η οικονομία και δημιουργήθηκε εισόδημα. Και αυτό είναι ένα δίδαγμα που πρέπει να μας πει κάτι. Και ελπίζω ότι τα μέλη αυτής τη Επιτροπής κάτι θα μάθουν από αυτό το μάθημα, καθώς ετοιμάζονται να γράψουν την εκθεσή τους. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, uh, Mr. Chairman, and uh, to all the Member of Parliament for having invited me here today. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που με καλέσατε σήμερα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μέχρι στιγμής. Βεβαίως, ε, εγώ θα μιλήσω για την ε, πολιτική του προπολισμού σε ένα εργαλείο για την οικονομική ανάκαμψη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να θυμόμαστε ότι η κατάσταση αυτή είναι πρωτοφανής γιατί η κρίση είναι η χειρότερη κρίση που έχουμε δει από την ύφεση του 1930 και δεν ξέραμε τότε τι έπρεπε να κάνουμε. Τώρα πειραματιζόμαστε με νέα εργαλεία και προσπαθούμε και να ανακάμψει η οικονομία και να δούμε πώς θα βγούμε από την κρίση. Αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ είναι ότι μαζί με την στρατηγική εξόδου πρέπει να έχουμε μια στρατηγική εισόδου προς περισσότερη ανάπτυξη πρώτα απ' όλα. Να σας υπενθυμίσω πως ε, έχουν εκραγεί τα ευρωπαϊκά δημόσια οικονομικά τελευταία χρόνια και έχουμε υψηλότερα χρέη και ελλείμματα που απειλούν το ρυθμό ανάπτυξης. Βλέπετε εδώ πέρα το δημόσιο χρέος ε, των 27 χωρών και της Ευρωζώνης. Ε, αυτά δεν είναι προβλέψεις. Είναι προβολές χωρίς να λάβουμε υπόψη ε, μέτρα που θα λάβουν οι χώρες για να συμμορφωθούν ε, με τα προβλήματα ειδικά του πληθυσμού που θα γερνάει. Όπως είπα, τα δημόσια ελλείμματα και η αρνητική ανάπτυξη. Έχει δείξει το Διεθνές Ζωνοματικό Ταμείο η εκτιμήση του πως μία μείωση ε, κατά 10% του δημοσίου χρέους ε, του ποσοστού με του δημοσίου χρέους ναι, οδηγεί σε μείωση της αιτής ανάπτυξης στα 0,2% λόγω και των υψηλότερων επιτοκίων και να σας επινομήσω εδώ πέρα πως η πρόβλεψη της ανάπτυξης ε, για την Ευρωζώνη μειώθηκε από 2% σε 1% από την Κομισιόν λόγω της κρίσης κατόπιν Έχουμε αυτό το οποίο έχουν πει Πατήγιο, Πορσόν και Ρίτσι που βρίσκουν αρνητικό και σημαντικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη επίπεδου σε στην ανάπτυξη με του χρέους σε υψηλά επίπεδα χρέους και για 15 χρόνια πριν από την κρίση ούτως ή άλλως με αυτό το αρνητικό σχετισμό στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Μπορούμε να βγούμε από την ε, κρίση μόνο με την αύξηση των επιτυχίων. Το θέμα είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό. Την αύξηση, με συγχωρείτε, της ανάπτυξης. Οπότε βλέπουμε τι γινόταν στο παρελθόν σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο και τη ΣΥΠΑ, ακόμα και αν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο από πλευράς πληθυσμού, είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπα. Τα στοιχεία αυτά είναι και σε ποσοστό και απόλυτα νούμερα και σε... στο ΑΕΠ είναι μεγαλύτερη από τις είπα. Τώρα πώς θα αυξηθεί η ανάπτυξη και ταυτόχρονα να διορθώσουμε το δημόσιο χρέος. Πρέπει να δούμε ποια είναι η δομή των δημοσίων δαπανών και το επίπεδο της ε, φορολογίας. Ο πληθυσμός που γερνάει θα αυξήσει τα δημόσια ελλείμματα στο μέλλον μέχρι ένα ποσοστό του 5% του ΑΕΠ ετησίως στην Ευρωζώνη εν μέρη λόγω των υψηλότερων δαπανών συντάξεων, λόγω των δαπανών υγείας επίσης. Τι θα κάνουμε τώρα με την αύξηση των δημοσίων δαπανών. Μπορούμε να αυξήσουμε τη φορολογία, αλλά ξέρουμε πως αυτό θα έχει αντίθετα αποτελέσματα αρνητικό αντίκτυπο στην ε, ανάπτυξη. Επίσης μπορούμε να κόψουμε τις δαπάνες, αλλά κάποιες δαπάνες έχουν ε, πολύ ισχυρή επίδραση στην ενίσχυση της ανάπτυξης αυτές που είναι έρευνα και ανάπτυξη, υποδομές και εκπαίδευση. Ποιε είναι λοιπόν οι στρατηγικέ εξόδου. Πρέπει να σφίξουν οι δημοσιονομικοί κανόνες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να αυξηθεί η αξιοπιστία του προπολογισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της δημόσια διοίκηση, να υπάρξουν δηλαδή κάποια στοιχεία που ε, θα μετράνε την απόδοση και όχι μόνο τις ε, δαπάνες, ε, αξιολόγηση της απόδοσης με συγκεκριμένους στόχους, επίσης να υπάρξουν συγκεκριμένα και πιστικά μέτρα μείωσης του στόχους, να, του κόστους, να αυξηθεί να αυξηθούν οι συμπράξει δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, να μεταρρυθμιστεί ο τομέα των συντάξεων και η αποτελεσματικότητα του τομέα τη υγεία. Αλλά εγώ θα επικεντρωθώ λίγο περισσότερο στο πώ ε, θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια στρατηγική ε, εισόδου για να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μέλλον. Το πώ θα έχουμε περισσότερου πόρου και καλύτερε προσπάθειε στην έρευνα και ανάπτυξη να δώσουν προτεραιότητα στι υποδομέ και με τα ρυθμίσεις φορολογικές που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη. Πώς θα έχουμε λοιπόν περισσότερη απόδοση της ε, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η κοινωνία γερνάει και δεν θα πρέπει έτσι να χάσουμε μια γενιά ολόκληρη λόγω της ε, κρίσης. Το να εξυγχρονίσουμε επίσης την αγορά εργασίας προ τον τομέα της ευελιξίας με ασφάλεια για να μπορούν οι άνθρωποι να αλλάζουν δουλειά με τις ε, ικανότητε που θα έχουν. Η αρχή επίσης ευελιξίας με ασφάλεια πρέπει να πάει χέρι με χέρι με τις απαραίτητε μεταρρυθμίσεις ε, για να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της ανεργίας. Και βεβαίω πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική αλλά αυτό σημαίνει πως θα έχουμε και ανακούφιση των συστημάτων κοινωνικής ε, πρόνοιας, ειδικά η συμμετοχή νέων γυναικών και γυναικών και των ηλικιωμένων θα γίνει μέσω μιας ενεργούς πολιτικής αγοράς εργασίας και ευελιξίας του χρόνου εργασίας. Επίσης ε, πρέπει να να ενισχυθούν τα συστήματα εκπαίδευση στην Ευρώπη και έτσι ώστε να βελτιώνουν συνεχώς δεξιότητε του οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι. Νέων καλύτεροι πόροι και περισσότεροι πόροι στην έρευνα και ανάπτυξη για να φτάσουμε το στόχο του 3% που θα ξοδεύεται στην έρευνα και ε, ανάπτυξη, κάτι το οποίο μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ της κοινότητας από 2,6 μέχρι 4,4% το να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα των πολιτικών δημοσιαστήριξης ε, έχει κρίσιμη σημασία για να εξοδεύονται καλύτερα τα ευρώ. Αυτό γίνεται μέσω καλύτερου συντονισμού των εθνικών πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης και με την ευρωπαϊκή με ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Επίσης, υποδομές. Τα επόμενα 10-15 χρόνια έχουμε μεγάλες ανάγκες υποδομών 3 εκατομμυρίων ευρώ. Οι στόχοι συμπεριλαμβάνουν ε, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ε, δυνατότητες παραγωγής ενέργειας ε, και ΑΠΕ. Ο περιβαλλοντικός τομέας, τα νερά, καταστροφή, κατασκευή με συγχωρείτε, αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τέλος, μεταρρύθμιση φορολογικού συστήματος πρέπει να γίνει πιο ίση συμμετοχή στο σύστημα, απλοποίηση του συστήματος, να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης, έτσι ώστε να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις και να είναι αυτές πιο βιώσιμες και αυτό θα συνεισφέρει σε μεγαλύτερα ωφέλη στην εσωτερική αγορά, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Thank Έχουμε και τον καθηγητή Μαρκ Χάλερμπεργκ, ο οποίος έγραψε ένα ενημερωτικό σημείωμα και νομίζω θα μπορέσουμε να βρούμε λίγα λεπτά να τον ακούσουμε. Νομίζω κάτι το οποίο είπατε βρίσκει αντίθετη κυρία Πέτιφορ. Οπότε θα μπορούσατε σε τρία λεπτά να συνοψίσετε τη θέση σας. Vielen Ας τα πω στα αγγλικά καλύτερα. Στο... Προφανώς δεν έχω το χρόνο να επισέλθω σε όλες τις λεπτομέρειες. Έχω μόνο δύο επιχειρήματα που θα ήθελα να σας διαμηνήσω. Πρώτον, αν ε, υπάρχει επιλογή ε, από την Ευρώπη, ε, μην ξεχνάτε τον τίτλο το δραματικό ότι βρισκόμαστε στα σταυροδρόμοι στην Ευρώπη. Ε, μπορούμε να δούμε τι έγινε σε άλλες ομοσπονδίες. Ε, φυσικά εμείς δεν είμαστε καθαρή ε, ομοσπονδία, αλλά μπορούμε να μάθουμε κάποια μαθήματα. Ε, μία δυνατότητα είναι να αναπτύξουμε μια πειθαρχία της αγοράς. Ε, οι αγοράς έχουν κακή φήμη σήμερα, το ξέρω αλλά θα εξακολουθήσω να ισχυρίζομαι ότι πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να συμβιώσουμε τις αγορές. Γιατί μας, οι αγορές μας δίνουν ε, τα χρήματα για τα ομόλογα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, να τις χρησιμοποιήσουμε τις αγορές αποτελεσματικά. Ε, είναι χρήσιμες οι αγορές, παρότι έχουν ατέλειες, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο τι μπορεί να κάνει τώρα για να ε, ενδυναμώσει την ε, πειθαρχία στις αγορές. Ε, Παραδείγματο χάρη στι ΗΠΑ τα ομόλογα ε, λειτουργήσαν σωστά ε, μέσα σε ένα πλαίσιο ε, πειθαρχίας αγοράς. Ε, εντάξει, ήταν σωστές οι τιμές. Ε, οι διάφοροι δήμοι και κυβερνήσεις, μιλάμε για τα ομόλογα των δήμων και των ε, ε, κοινοτήτων, λειτουργήσαν σωστά. Αν δείτε το, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η βασική πρόκληση είναι να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί πρόληψης, ούτως ώστε να υπάρχει περισσότερη ενημέρωση από τις αγορές και περισσότερη ενημέρωση για τον πληθυσμό αυτό θα συμπληρώσει αυτό που κάνουν οι αγορές και θα στείλει το σωστό μήνυμα για τις αγορές. Αν κοιτάξετε τι συμβαίνει, πολύ λίγοι άνθρωποι καταλαβαίνουν τα μηνύματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ε, συγκρίναμε την Κομισιόν και, την, και το Συμβούλιο ως προς τις συστάσεις τους. Ε, το Συμβούλιο νομίζω κάποια στιγμή αποδυνάμωσε ε, τις συστάσεις της ε, Κομισιόν. Υπήρχε μια σύγκρουση δηλαδή. Μια εναλλακτική λύση είναι χαμηλότερη πειθαρχία στις αγορές. Ε, τότε όμως θα πρέπει να έχουμε μια κάποια πολιτική ολοκλήρωση το δεύτερο τμήμα του εγγράφου λέει «Κοιτάξτε τη Βραζιλία, κοιτάξτε, αν θέλετε να εμπνευστείτε για κάποιο μοντέλο, κοιτάξτε». Ε, πριν από το 2000 θεωρούσαμε ότι ήταν μια σχετική καταστροφή η Βραζιλία, αλλά έγιναν διάφορες μεταρρυθμίσεις, ε, ε, διαπραγματεύσεις, ε, σε κεντρικό επίπεδο, οι οποίες παρακολουθούνταν και δημοσιεύονταν ε, υπήρχαν σε κάθε πολιτεία ε, δημοσιονομικά συμβούλια, ε, παρακολούθησε το τι έκανε η κεντρική κυβέρνηση. Αυτό το συζητάμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αν οι πολιτείες δεν ε, συμμορφώνονται, δύο πράγματα μπορούν να γίνουν. Ε, τότε οι πιστώσεις από την κεντρική κυβέρνηση μειώνονται. Έχει συμβεί αυτό στην Βραζιλία. Και το δεύτερο, που θα ήταν πολύ ριζοσπαστικό για την Ευρώπη, είναι ότι αν συνεχίσει αν συνεχίσουν κάποιοι πολιτικοί ας πούμε, να ξεπερνούν κάποια όρια, μπορούν να καταλήξουν στη φυλακή. Αυτό είναι πάρα πολύ εξικέλευθο, αλλά έγινε σε ορισμένε περιπτώσει, κυρίω δήμαρχοι στη Βραζιλία κατέληξαν στη φυλακή. Ε, ίσως είναι υπερβολικά ακραίο. Αλλά η ιδέα είναι ότι υπάρχει ένα σύστημα όπου ε, έγιναν διάφορες διασώσεις. Ε, κάποια στιγμή έπρεπε να σταματήσει. Το θέμα είναι τι αλλαγές πολιτικές έπρεπε να γίνουν για να σταματήσει αυτή η ιστορία. Αυτά ευχαριστώ και τον χρόνο. Uh, και τώρα ερωτήσεις. Κυρία Άλβαρες είναι η πρώτη. Ο κύριος Βάγκον, Βόγγελ. Και ο Πασκάλ δεν θέλει να κάνει ερωτήσεις, έτσι. Όχι, δεν θέλει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Σήμερα το πρωί εμείς εξετάσαμε τις δυνατότητες για έξοδο από την τωρινή κρίση αλλά και για να αποφύγουμε να ξαναμπούμε σε κρίση. Κάποιος είπε ότι αρκεί και μόνο να εφαρμόσουμε τους τωρινούς κανόνες. Όμως μας θύμισαν ότι χώρες όπως η Ισπανία αλλά και άλλες εφαρμόστηκαν όλοι οι κανόνες αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη Ευρώπη. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πέρες. Ε, τι σκέφτεται για την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου αντίστοιχου με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πώς θα έπρεπε να πρικοδοτηθεί, ποιος θα ήταν ο ρόλος του και πώς θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα Ταμείο Εγγύσεων και Καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν ξεκίνησε η ακρόαση, η ακρόαση μάλλον, μιλούσαμε για χρηματοπιστωτικό έλεγχο και χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς. Τώρα φτάσαμε σε μια στιγμή όπου η χρηματοπιστωτική κρίση έγινε και κοινωνική κρίση. Φυσικά οι ομιλητές του πάνελ δεν μπορούν να κρίνουν πόσο πόση υποστήριξη από τους λαούς της Ευρώπης έχουν τα νέα εργαλεία. Τι είναι έτοιμοι οι ευρωπαϊκοί λαοί να κάνουν. Το ερώτημα υπάρχει βέβαια. Ορισμένοι από τους ομιλητές του προηγούμενου πάνελ είπαν ότι υπάρχουν κάποιες ε, λαϊκιστικές πολιτικές, κάποιες δημαγωγικές πολιτικές που μπορεί να αυξηθούν λόγω της κρίσης ή μπορεί να τις προκαλέσει η κρίση. Και εγώ συμμερίζομαι αυτό το φόβο. Και όταν μιλούσαμε για την ελληνική κρίση και ακούσαμε την αισιόδοξη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν μπορούμε να μη σκεφτούμε τις εικόνες που βλέπουμε κάθε μέρα στον τύπο. Βλέπουμε την απροθυμία του λαού να καταπιεί αυτό το πικρό χάπι. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για αυτά τα σχόλια που κάνω. Και θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία του πάνελ που μίλησε για την Ιαπωνία. Εγώ πρόσφατα επισκέφθηκα αυτή τη χώρα και μίλησα στον πρώην Υπουργό Οικονομικών της Ιαπωνίας, ο οποίος μας ρώτησε πώς και δεν αναλύσαμε και δεν μάθαμε κάτι από την ε, Ιαπωνέζικη εμπειρία. Γιατί δεν τη μελετήσαμε αυτή την κρίση. Γιατί δεν τη μελετήσαμε την περίπτωση Ιαπωνία. Ιαπωνίας. Ευχαριστώ. Για το θέμα του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, ήδη σήμερα το πρωί ακούστηκαν με δικέ ιδέες. Τώρα ως εκτελεστικός διευθυντής ε, του Νομισματικού Ταμείου εγώ θα ήθελα να αναφέρω δύο στοιχεία που θεωρώ ότι είναι αδιαμφισβήτητα για να δημιουργήσει το Eurogroup η Ευρωμάδα έναν μηχανισμό επικουρίας, έναν μηχανισμό αρρωγής μέσα, δημιουργώντας ένα κοινό ταμείο. Το βασικό λάθος θα ήταν να ονομαστεί αντίστοιχα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Σας θυμίζω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε περίπτωση που μία χώρα της ζώνης του ευρώ πάει θα συμφωνήσει γύρω από ένα πρόγραμμα και θα χρηματοδοτήσει κατά μεγαλύτερο μέρος με τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όμως στη διαχείριση αυτού του χρήματος θα συμμετέχουν όλοι όσοι βρίσκονται, όλες οι χώρες εκείνες που βρίσκονται στην διεύθυνση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μετά Όλα εξαρτώνται από το πώς παρακολουθείτε ή παρακολουθούνται οι εξελίξεις στην ενδιαφερόμενη χώρα και το πώς αυτή η χώρα σε περίπτωση που δεν εκπληρώσει τους στόχους της ή κάνει κάποια παράβαση να βρεθεί χωρίς βοήθεια. Σε περίπτωση που μία χώρα ευρωπαϊκή βρεθεί υπό τον έλεγχο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε περίπτωση που δεν θα εκπλήρωνε τους όρους της θα βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και την απόφαση θα την, θα την έπαιρνε το Διευθυντικό Όργανο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Λοιπόν, ποιος θα χρηματοδοτήσει και πώς θα μπορούσε κανείς να διαχειριστεί το πρόγραμμα σε συνεργασία με την ενδιαφερόμενη χώρα είναι ουσιαστικό αυτό να γίνεται μέσα στη ζώνη ευρώ με τη χορήγηση μίας οικονομικής ενίσχυσης την οποία θα ελέγχει η Ευρωμάδα. Τώρα, εδώ μιλάμε για ενίσχυση, για βοήθεια. Αν υποθέσουμε τώρα ότι μια χώρα πάει, προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πώς χρηματοδοτείται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τα αποθέματα των κεντρικών τραπεζών των διαφόρων χωρών που τροφοδοτούν το Ταμείο, είτε Διεθνές Τράπεζες. Λοιπόν, το, το κονδύλι επενδύεται εκεί με τη μία αγοράς και δίνεται μία αποζημίωση στη χώρα προέλευσης. Και εμείς μπορούμε μόνο στο διευθυντή του να ρωτήσουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, και πώς έχει η εποπτεία έναντι της ενδιαφερόμενης χώρας. Πρόκειται για ένα απλό ευέλικτο σύστημα, κάτι αντίστοιχο θα έπρεπε να λειτουργεί και στην Ευρώπη. Θα έπρεπε λοιπόν, επειδή πρόκειται για έκτακτες καταστάσεις, να έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα ενίσχυσης, κατεπίγουσας ενίσχυσης στην ενδιαφερόμενη χώρα. Για, τώρα, ποιο είναι το ιδανικό ενός προγράμματος του, Διεθνές, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή, χορηγείται με το κονδύλι, αλλά δεν δίνεται στη χώρα, δεν το διαθέτει η χώρα. Το 60 προσέφυγε η Ισπανία στο Διεθνές νομισματικό ταμείο. Αλλά δεν πήρε δολάριο. Από μόνη της μπόρεσε να ξεπεράσει την κατάσταση. Τώρα για το Ταμείο Καταθέσεων και Εγγύσεων. Η Ισπανία έχει μία εμπειρία και αυτό λόγω της οικονομικής κρίσης ε, στα τέλη του 70 και αρχές 80. Αυτό το Ταμείο Καταθέσεων και Εγγύσεων είναι κάτι το εντελώς ιδιωτικό δηλαδή είναι οι τράπεζες ε, που συνεισφέρουν και πρικοδοτείται απριόρι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε κρίση μιας τράπεζας όπου πρέπει βιαστικά να χρηματοδοτήσουμε αυτό το ταμείο. Και ε, η λειτουργία του είναι διπλή, δηλαδή είναι ένα ταμείο εγγύσεων αλλά αποτελεί και μέσω βοήθειας μίας τράπεζας που περνάει κρίση. Πώς θα μπορούσαμε τώρα να το εξομοιώσουμε αυτό με ένα ασφαλιστικό πριμ. Ένα ασφαλιστικό πριμ μπορεί να είναι πιο φτηνό και πιο αποτελεσματικό. Όταν οι διαχειριστές του Ταμείου αποφασίσουν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η τράπεζα, να ορθοποδήσει αντί να κλείσει η τράπεζα, να φαλυρίσει και να αποζημιωθούν όλοι οι καταθέτες που είναι πολύ πιο πολύπλοκο. Αυτό είναι σαφώς πιο εύκολο. Για να σας απαντήσω σε αυτό το οποίο είπατε. Ε, πολύ πατρονάρισμα υπάρχει για το λαϊκισμό. Δικαίως οι άνθρωποι δυσανασχετούν όταν πρέπει να υπομισθούν το βάρος ε, της προσαρμογής. Η κρίση στην Ευρωζώνη όπως είπε ένας δημοσιογράφος των ε, Financial Times, είναι θέμα ιδιωτικής έλλειψης επιθαρχίας, αλλά την πληρώνει ο δημόσιος τομέας. και υπάρχουν και όρια στο τι μπορεί να γίνει πολιτικά. Δόξα τω Θεώ που ζούμε σε δημοκρατία. Σε δημοκρατίες στις οποίες οι άνθρωποι δεν τα ανέχονται αυτά τα πράγματα. Και αυτοί που χαράζουν την πολιτική δεν πρέπει να λυπούνται για το ότι ζούμε σε δημοκρατίες. Πρέπει να είναι θετικοί. Στην Ιαπωνία, ε, για το δόνοτου, ελπίζω πως ε, εάν αρχίσει να στείνει νομισματικό ταμείο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην βασιστεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει διαρθρωτικά προβλήματα. Το μεγαλύτερο από τα οποία είναι ότι δεν έχει την εξουσία ή δεν ασκεί την εξουσία να πειθαρχήσει τις χώρες τις πλεονασματικές και όχι μόνο τις ελληματικές. Αφορά μόνο τις πλεονασματικές χώρες και άρα στην παγκόσμια οικονομία έχουμε πάρα μεγα, πολύ μεγάλες ανισορροπίες π.χ. μεταξύ ΙΠΑ και Κίνας και το Διεθνές Ταμείο δεν έχει κάνει τίποτα για να διορθώσει αυτές τις ανισορροπίες. Οπότε, εάν να στήσουμε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, πρέπει να είναι διατεθειμένο να αντιμετωπίσει τη Γερμανία και το πλεόνασμά της. Δεν είμαι σίγουρη βεβαίω αν θα το δεχτούν αυτό οι Γερμανοί, αλλά θα είναι ένα από τα μεγάλα καθήκοντά του. Να πω τώρα στην, για την Ιαπωνία. Ναι, δεν έχουμε διδαχτεί από την Ιαπωνία. Θεωρούμε ότι η Ιαπωνία είναι κάτι περιφερειακό στην παγκόσμια οικονομία. Αλλά η Ιαπωνία πέρασε ακριβώς αυτό το οποίο περνάμε εμείς τώρα. 1987 μείωσε τα επιτόκια της αντιδρώντας την οικονομική κρίση, την κρίση στα ομόλογα του 1997 Μετά δημιουργήθηκε μια φούσκα των ακινήτων που εξεράγει και 20 χρόνια μετά ακόμα έσκασε η φούσκα. Ακόμα δεν έχει συνέλθει η Απονία το σκάσιμο αυτής της φούσκας. Για να σα το πω ε, εδώ να το καταλάβετε. Άρχισαν να πέφτουν πριν από 20 χρόνια και εξακολουθούν να πέφτουν οι τιμές των σπιτιών στην Ιαπωνία. Φανταστείτε να συμβεί κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Οπότε νομίζω ότι δεν έχουμε διδαχθεί ακόμα ε, εγώ ανησυχώ, παρακολουθώ τους ε, βασικούς δείκτες του πληθωρισμού στην Ιαπωνία και έπεσαν πάλι αυτό το μήνα και νομίζω πως οι Γερμανοί ανησυχούν πάρα πολύ για το θέμα του πληθωρισμού και δεν αντιλαμβάνονται πλήρως την ε, πολύ πιο τρομακτική πιθανότητα του αποπληθωρισμού όπου ο κόσμος απομοχλεύει, όπου ο ιδιωτικός τομέας απομοχλεύει μαζικά και μετά έρχονται εδώ πέρα οι οικονομολόγοι και μας λένε πως ο δημόσιος τομέας πρέπει να κάνει το ίδιο. Και ο συνδυασμός ε, ιδιωτικής και δημόσιας απομόχλευσης θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποπληθωρισμό. Είναι τρομακτικό αυτό. Φοβάμαι πως οι οικονομολόγοι μας δεν, ε, δεν το έχουν ε, συλλάβει ειδικά στη Γερμανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε, να επανέλθω στην Ιαπωνία. Είπατε πως δεν έχουμε βγάλει τα σωστά συμπεράσματα. Και λέτε, νομίζω, την τελευταία δεκαετία έχουν αντλήσει οι Ιάπωνες οι ίδιοι τα τα διδάγματά τους και έριξαν χρήμα στην οικονομία όσο μπορούσαν. Δηλαδή το συνολικό χρέος είναι πόσο, 250%. Τέλος πάντων, εφόσον αναφερθήκατε στο θέμα του πληθωρισμού, γίνεται λόγο στην Αμερική για το ότι ε, δεν έχουν επίσημο στόχο ούτως ή άλλως, αλλά λένε ίσως θα μπορούσαν να πάνε κάπου στο 4%. Λέγοντα πως ίσως θα έπρεπε να το ακολουθήσει αυτό και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αντί να είναι κάτω και κοντά στο 2% να είναι πιο ευέλικτη. Και να πούνε πως ίσως για κάποια περίοδο να σκεφτούμε το 3-4 κτλ. Πρώτο ερώτημα, τι άποψη έχετε γι' αυτό, για αυτή τη σύσταση. Δεύτερον, όποια και να είναι η σύσταση, μήπως δεν θεωρείτε πως ούτως ή άλλως στο τέλος θα έχουμε μεγάλο πληθωρισμό δεδομένων των ε, τεράστιων επιπέδων του χρέους. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν οι περισσότερες χώρες να ξεφύγουν από αυτό. Και ήδη έχω την αίσθηση υποκειμενική πως ε, η Αμερική θα προσπαθήσει να λύσει αυτό το μέρος του προβλήματος να αρχίζουν να τυπώνει χρήμα. Επιταχύνοντας ε, την, την διαδικασία αυτή μιλάνε για ισχυρό δολάριο, αλλά de facto τους ενδιαφέρει ε, το ασθενές δολάριο για τις εξαγωγές τους. Και βεβαίω η Κομισιόν μόλις δημοσίευσε στρατηγική του 2020. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί. Πάμε σωστή κατεύθυνση ή είναι έτσι, από αυτά τα, τα έγγραφα που δεν ε, θα μας ε, βοηθήσουν να, κάνουμε αυτά που πρέπει τα επόμενα δέκα χρόνια. Well, you very much. Let me start... ε, σας ευχαριστώ να ξεκινήσω με λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό ε, Ταμείο και τις εγγυήσεις στις ε, καταθέσεις η άποψή μου. Δεν έχω άποψη εγώ για το πώς πρέπει να οικοδομηθούν αυτοί οι μηχανισμοί. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξει ένας πιο συμμετρικός ε, μηχανισμός όπως είπε η κυρία Πέτιφορ αν και το ζήτημα εντός ε, της Ευρώπης δεν είναι πάντα η χρηματοδότηση ξένων ε, ανισορροπιών, γιατί είμαστε σε Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Για μένα είναι πάντα δύσκολο μετά να φανταστώ μια ευρωζώνη ή ένα το πώ ε, θα έχουμε μηχανισμό ενιαίου νομίσματος χωρίς να έχουμε με ενιαία αγορά. Πρέπει να θυμόμαστε την σταδιακή οικοδόμηση της Ευρώπης. Πρέπει να θυμόμαστε πως με βάση την αγορά σκεφτήκαμε πω πρέπει να έχουμε και ενιαίο νόμισμα. Τούτου λεχθέντος συμφωνώ πως ε, και ε, οι Ιαπωνέζοι έμαθαν πως πώς πρέπει να διαχειριστούν την ανάπτυξη, ακόμα και με επιτόκια μηδέν. Και προσπαθώντας ε, να παλέψουν με ένα χρέος, με ένα έλλειμμα, με συγχωρείτε, γύρω στο 7%. Είναι χαμηλός ο, ο πράγματι και νομίζω γενικά στην Ευρωζώνη είμαστε σε ένα αποπληθωριστικό περιβάλλον. Οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος αυξημένου πληθωρισμού. Η πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να διευρύνουμε το εύρος του στόχου του πληθωρισμού δεν μας χρησιμεύει αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως, εάν ήμασταν σε μια κατάσταση πληθωριστικών πιέσεων, είναι δύσκολο να θέσουμε τον πληθωρισμό υπό έλεγχο όταν αυξάνονται οι προσδοκίες, οι πληθωριστικές. Ε, είναι δύσκολο λοιπόν να πούμε πως είναι χρήσιμη αυτή η πρόταση. Τέλος, για το ασθενές δολάριο, δεν νομίζω πως ε, ούτε και η κυβέρνηση Ομπάμα δεν μπορεί να αποφασίσει ποια θα είναι η ισοτιμία του δολαρίου. Υπάρχουν τεράστιες ε, κινήσεις ε, κεφαλαίων ε, γύρω από την Ιφίλιο και δεν μπορούν να τα ελέγξουν αυτά. Να πω, ο κύριος Παολάτση ανέφερε κάτι πολύ φοβερό, ότι οι κυβερνήσεις, ακόμα και οι κυβέρνηση των ΗΠΑ, δεν έχουν αυτονομία στην πολιτική τους. Και νομίζω πως αυτό άρχισαν να το καταλαβαίνουν ε, οι άνθρωποι. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτές τις κρίσεις προς το συμφέρον των ανθρώπων. Που δεν θα είναι πράγματα αποδεκτά σε ανθρώπους ε, όπως εμείς. Πρέπει και να επιτρέπουμε στον ε, τομέα των χρηματαγορών να κάνει ό,τι θέλει στον, στον κόσμο. Οπότε επανερχόμαστε στην κινητικότητα του κεφαλαίου και στον έλεγχο του κεφαλαίου που είναι κάτι που κανείς δεν θέλει αν και βλέπω πω το Διεθνές Νομοθετικό Ταμείο αρχίζει να λέει πω πρέπει να συζητήσουμε ελέγχου του κεφαλαίου, κάτι το οποίο με ενθαρρύνει μετά από χρόνια συνεργασία με το Διεθνές Νομοθετικό Ταμείο, το οποίο αποτυγχάνει να προβλέψει, απέτυχε να προβλέψει την κρίση τη Λατινική Αμερική της Νοτιοανατολικής Ασίας και αυτή την κρίση. Και το γνώριζαν ε, λόγω λανθασμένη οικονομική πολιτική Είχε στην Ιαπωνία. Δεν είμαι ειδική. Αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να πω στον Πρόεδρο, υπάρχει μία λεπτή ακολουθία που πρέπει να ακολουθεί χρησιμοποιώντας και δημοσιονομικά κίνητρα και αν η σειρά αυτή δεν γίνει σωστά όπως έγινε στην Ιαπωνία καταλήγουμε με αυτό το οποίο είπε ο φτάνουμε στα άκρα και ε, ήταν πάρα πολύ αργοί δεν αντιλήφθηκαν ε, πως ε, λάμβανε χώρα η διαδικασία αυτή απομόχλευσης και τον Ιούλιο αύξησε τα επιτόκια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Διανόητο, Η δε Κεντρική Τράπεζα τη Ιαπωνία είχε κάνει παρόμοια λάθη. Και άρχισαν οι άνθρωποι να αποταμιεύουν, να τα βάζουν κατά το στρώμα. Δεν επενδύουν. Μπορεί και εμείς να φτάσουμε στην ίδια κατάσταση. Εγώ φοβάμαι πως κάποιες από τις ιδεολογικές προσεγγίσεις εδώ πέρα μας δυσκολεύουν να σκεφτούμε με καινοτόμο τρόπο, διαφορετικά από την Ιαπωνία. Περβάνος Μπερές, η συγγήτριά μας, είναι η τελευταία. Θέλω να κάνετε μία ερώτηση όχι. Έχω εγώ μία μικρή ερώτηση για τις ερωτήσεις του Πρόεδρου. Ε, με τις οποίες ε, συμφωνώ η περίπτωση της Ιαπωνίας μας δείχνει ξεκάθαρα το πόσο η εργοπορία και ο δισταγμός ε, στη λήψη αποφάσεων οδήγησε σε 30 χρόνια χαμηλής ανάπτυξης με αποτέλεσμα ένα επίπεδο χρέους το οποίο είναι τραγικό, είναι πολύ υψηλότερο από αυτό το οποίο θα είχε δημιουργηθεί από οποιοδήποτε πρόγραμμα κινήτρου. ενώ η Απονία έχει πολύ υψηλό επίπεδο αποταμιεύσεων οπότε μπορεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί με τρόπο που δεν μπορεί να το κάνει κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τώρα τον κίνδυνο πληθωρισμού και σήμερα η ανησυχία θα πρέπει να είναι ανάπτυξη και απασχόληση. Ο πληθωρισμός δεν είναι στο ραντεβού, ούτε τον περιμένουμε. Σίγουρα θα επανέλθουμε σε καταστάσεις με πληθωριστική ε, απειλή. Αλλά τελικά αν κάτι μπορεί να κάνει η Κεντρική Τράπεζα είναι να παρουσιάζει ε, προγράμματα που να διαφυλάσσουν τη σταθερότητα των τιμών. Αυτό όμως το οποίο δεν μπορεί να κάνει καμία τράπεζα στον κόσμο είναι να ελέγξει τον αποπληθωρισμό. Λοιπόν και για λόγους χρονοδιαγράμματος και για να κάνουμε αυτό το οποίο ξέρουμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε την κεντρική τράπεζα να ε, κάνει ενέσεις χρήματος στην αγορά ούτως ώστε να συνεχίσει να είναι γενεσιουργός απασχόλησης ε, ένα γρήγορο σχόλιο για τα πλεονάσματα, τη Γερμανία και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών πληρωμών. Όταν η Κίνα έχει ένα πλεόνασμα στο ισοζύγιο του τρεχουσών πληρωμών, μπορεί το νόμισμα να αναβαθμιστεί. Στη Γερμανία όμως είναι πολύ πιο δύσκολο, ε, λόγω της νομισματικής ένωσης. Αυτή η συζήτηση είναι πώς τελικά θα μειώσουμε την ανταγωνιστικότητα στη Γερμανία, ούτω ώστε να είναι ανταγωνιστικέ οι τιμέ του. Αν κοιτάξετε τα πράγματα από την σκοπιά των Γερμανών, ε, το, η προοπτική για ανάπτυξη της Γερμανίας είναι 1%. Είναι χαμηλή. Το θέμα είναι, και αυτό που την ανησυχεί τη Γερμανία, είναι πώς θα το αυξήσει. Ε, επίσης, ο πληθωρισμός είναι γύρω στο 4%. Αυτό συνδέεται με την κρίση όμω. Αλλά οι μεταρρυθμίσει που χρειάζονται είναι ε, μεταρρυθμίσει για να αυξηθεί η ανάπτυξη. Είναι μια γυράσκουσα επίση κοινωνία που έχει πάρα πολλά προβλήματα ε, με του ε, μισθού κτλ. Ε, και επίση υπάρχουν προβλήματα με τα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τροχουσών πληρωμών. Ω συνήθω υπερβάλλουν στο τελευταίο λόγο. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους με τους προσκεκλημένους. Πραγματικά δεν θα το αντέξω να μην κάνω μερικά σχόλια για το τελευταίο σχόλιο, για το τελευταίο πάνελ. Τώρα κύριε Πέρε για, για, για τις αρμοδιότητες ε, της Κεντρικής Τράπεζας, μα το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι η συνθήκη δεν εφαρμόζεται και γι' αυτό. Εγώ από την αρχή πραγματικά πάλεψα να έχουμε μια πραγματική εφαρμογή της συνθήκης. Εγώ το είχα πει πάντα ότι όταν θα είχαμε πια τη σταθερότητα των τιμών η νομισματική πολιτική θα πρέπει να συμβάλλει όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 στην ολοκλήρωση των άλλων πολιτικών της Ένωσης. Αλλά δεν υδρώνει το αυτή κανενός για την Κεντρική Τράπεζα και λένε ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να πληρεί πολλούς ε, στόχους, μόνο έναν πρέπει να εξυπηρετεί. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε. Και δεν νομίζω ότι η κρίση τελικά αλλάζει την αντίληψη που έχει η ίδια η τράπεζα για το πώς ε, ερμηνεύει την εντολή της. Τώρα για τον κύριο Μπλανσάγ σχετικά με τον πληθωρισμό και το είπε και ο Στροσκάν εχθές ε, λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος του αποπληθωρισμού που είναι πολύ ε, σημαντικότερος. Οι ε, ονομαστικοί μισθοί στην Γερμανία μειώθηκαν κατά 3,6 το 2009, κάτι το απίθανο, δεν έχει συμβεί ποτέ. Το να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τον πληθωρισμό τελικά ίσως να δείχνει ότι δεν θα πρέπει να επανέλθουμε στην αφετηρία αλλά να προχωρήσουμε. Και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπλανσάρη είναι σωστό για να το δούμε πιο κοντά. Τώρα για την ε, Ιαπωνία. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε το σχέδιο ανάκαμψης στο τραπέζι είπαμε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχουν προοπτικές ανάκαμψης το 2011 και ότι είχαμε το ρίσκο να μπούμε σε μια στρατηγική Ιαπωνέζικου στυλ. Αλλά κανένας δεν κατάφερε να ηρεμήσει αυτή την ανησυχία. Τώρα δεν είναι ένα θέμα στυλ, αλλά το είπε και ένας άλλος συνάδελφος. Σε αυτές ε, τις ε, ακροάσεις ε, πολλές φορές ε, ξεχωρίζω τον έναν ή τον άλλον ομιλητή αυτή αυτήν εδώ την ακρόαση δεν μου συνέβη κάτι τέτοιο όλοι οι ομιλητές ήταν πάρα πάρα πολύ καλοί είχαμε μια συζήτηση ιδιαίτερα πυκνή ιδιαίτερα περιεκτική υπάρχει ακόμη ένα σωρό δουλειά σίγουρα δεν μας αρκεί μόνο αυτό για να βγούμε από τη γενική αταξία. Η διάρθρωση μεταξύ των δύο πάνελ ήταν πολύ εμπλουτιστική. Εγώ πραγματικά έχω έμονη ιδέα με το θέμα της οικονομικής ε, διακυβέρνησης, ε, ίσως γιατί είμαι Γαλλίδα σοσιαλίστρια. Αλλά βλέπω ότι η Ιαπωνία, η Αμερική έχουν μια οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό δεν τους ε, ωφέλησε στο να βγουν από την κρίση. Το θέμα είναι το πώς χρησιμοποιεί κανείς το δημοσιονομικό μέσο για να βγει από τις δυσκολίες. Και ένα άλλο, ε, το οποίο ελπίζω να με υποστηρίξουν ε, οι συνάδελφοι στην έκθεσή μου είναι το να μπορέσουμε να δούμε τον συνδυασμό της δημόσιας και της ιδιωτικής επένδυσης γιατί αλλιώς δεν βγαίνουμε από την κρίση και υπάρχει και ένας κίνδυνος σημαντικότατος για τη δημοκρατία μας άμα δεν βγούμε από αυτή την κρίση. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργό ο κύριος Παπανδρέου, ήταν καταπληκτικό για μας ε, να τον έχουμε μαζί μας σήμερα το πρωί. Αυτό το οποίο μας είπε για το τι θα έπρεπε και ποια θα μπορούσε να είναι η αντίδραση της Κομισιόν για την ευελιξία του ε, Συμφώνου Σταθερότητας. Την ευελιξία ο καθένας να την κάνει ό,τι θέλει και μετά ο Θεός ε, να παρέμβει άμα χρειαστεί. Ε, αυτό δεν είναι λύση. Σας ευχαριστώ πάντως ε, για τις τοποθετήσεις σας.